Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους. Παραλαμβάνω. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα αρχίσουμε την συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και όπως ήθιστε πρώτο θέμα είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Το σχέδιο το έχετε και προτείνω την εξής αλλαγή μία μόνο το σημείο 8 εισηγητής Χόπ για τα εγκληματολογικά εργαστήρια αυτό το θέμα λοιπόν προτείνω να το συζητήσουμε σαν πρώτο θέμα διότι ο εισηγητής θα πάει στη συνδιάσκεψη των προέδρων των πολιτικών ομάδων που λαμβάνει η χώρα σήμερα οπότε αν δεν υπάρχει αντίρρηση προτείνω το σημείο 8 να γίνει πρώτο θέμα συζήτηση σήμερα και μετά στις ανακοινώσεις του Προέδρου θα ήθελα να σας ζητήσω να εγκρίνετε τους εξής εισηγητές που αποφάσισαν συντονιστές Μακοβέι, σύστημα Eurodac για τη σύγκριση δακτυλικών αποτυπωμάτων των τρίτων χωρών ή α, απάτριδων ή απάτριδων. Μετά τρίτες χώρες με τις οποίες θα συνάψει ε, συμφωνίες η Ευρωπόλ. Ναι, ο κύριος... και γι' αυτό αυτά είναι οι δύο εισηγητέ, του οποίου αποφάσισαν συντονιστέ επί τη διαδικασία. Μάλιστα, καλημέρα πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι τι στις 13 Οκτωβρίου έγινε μια ενημέρωση και παρουσίαση την περασμένη Τρίτη στο Λονδίνο για εκρηκτικά, υγρά εκρηκτικά. Ε, είχαμε πάρει όλη πρόσκληση νομίζω όλα τα μέλη αυτής της Επιτροπής πήραμε τη σχετική πρόσκληση την 1η Οκτωβρίου οπότε προσπάθησα, ενδιαφέρθηκα, ε, προσπάθησα να βάλω το όνομά μου στον κατάλογο, αλλά τελικά είδα ότι η καταληκτική προθεσμία ήταν 8 Σεπτεμβρίου. Πώς μπορούμε να πάμε ε, και να δηλώσουμε συμμετοχή με ημερομηνία με προθεσμία 8 Σεπτεμβρίου όταν παίρνουμε την πρόσκληση 1 Οκτωβρίου. Μπορείτε να, το, να μου το εξηγήσετε αυτό, Πρόεδρος. Κοιτάξτε με κάθε σεβασμό, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι η πρόσκληση με τις προσκλήσεις ασχολήθηκε η Βρετανική κυβέρνηση. Εκείνη έστειλε σε κάποια μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φαντάζομαι πρόσκληση για το ε, σεμινάριο αυτό, για την παρουσίαση αυτή για τα υγρά, για εκρηκτικά, αλλά τη διαδικασία ακριβώ δεν ξέρω, δεν την ξέρω, εγώ δεν πήγα προσωπικά, δεν ξέρω αν υπάρχει κανείς άλλο στην αίθουσα που να έχει περαιτέρω πληροφορίες. Πάντως αναλαμβάνω να σας δώσω πλήρες ε, πληροφορίες για το τι συνέβη και πού συνέβη το λάθος τελικά. Γιατί νομίζω ότι βεβαίω σας οφείλεται μια απάντηση ο κύριος Κοέλιο. Από ό,τι θυμάμαι η πρώτη πρόσκληση ήρθε στην ώρα της αλλά η δεύτερη πρόσκληση αν θέλετε υπενθύμηση για τη συνάντηση αυτή έσταλει μετά το τέλος της προθεσμίας. Ούτε και εγώ πήγα στην επίδειξη αυτή αλλά ίσως αν κάποιος από την Επιτροπή μας πήγε να μπορέσει να μας ενημερώσει μελλοντικά πρόεδρος το σημειώνουμε και θα σας δώσουμε πράγματι τις πληροφορίες οι οποίες σας οφείλονται Λοιπόν, ας προχωρήσουμε με το σημείο 8 όπως είπαμε. Απόφαση πλαίσιο για τη διατήρηση της ασφάλειας των πληροφοριών όταν πρόκειται για σημαντικά προσωπικά δεδομένα όπως παραδείγματος χάρη στοιχεία DNA και δακτυλικά αποτυπώματα. ότι ε, είχαν υποβληθεί κάποια σχόλια, ε, ελήφθησαν γραπτές απαντήσεις από τη Σουηδική Προεδρία το, ε, το Κοινοβούλιο πρέπει να απαντήσει μέχρι τις 26 Νοεμβρίου I'm so sorry. I'm Uh, Επαναλαμβάνω. Πρόκειται για μια πρόταση τρίτου πυλώνα που μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση ισχύ τη συνθήκη της Λισαβόνα και αν δεν δημοσιευθεί έγκαιρα στην επίσημη εφημερίδα θα πρέπει να επανυποβληθεί ε, μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης. Ο εισηγητής είναι ο κ. Κέρκχοπ, ο οποίος έχει και το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Στο Ηνωμένο Βασιλείο έχουμε ένα... λέμε ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην βάλουμε το αμάξι μπροστά το άλογο να μην κάνουμε προθύστερα. Ε, αυτό συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ε, τα χρονοπρογράμματα που ορίστηκαν εδώ είναι για τους περισσότερους από εμά απαράδεκτα και γι' αυτό δηλώνω ήδη από την αρχή ότι μας βάζουν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Πρόκειται για μια απόφαση πλαίσιο μετά το Συμβούλιο των Υπουργών στις 9 Οκτωβρίου και κάπου στην αιτιολογική έκθεση λέγεται εκτιμώντας, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με συγχωρείτε, ε, ε, αυτό είναι πράγματι προθήσεις του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει γνωμοδοτήσει. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες για τη συνθήκη της Λισαβόνας και για το ότι αργότερα θα έχουμε περισσότερες εξουσίες αν θέλετε. Δεν το συζητώ αυτό, αλλά εκείνο που θα ήθελα να πω ότι αυτό που συζητούμε σήμερα είναι ελπίζω απλώς πρόδρομος μιας μελλοντικής ε, πρότασης την οποία θα συζητήσουμε εκτενέστερα. Ελπίζω δηλαδή να ξανασυνασχοληθούμε με το θέμα αργότερα όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει ε, τη δυνατότητα να εκφραστεί για το γενικότερο πλαίσιο για τη χρήση των πληροφοριών και τα λοιπά που είναι σοβαρά θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν. Δεν μιλούμε όμως για αυτά αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή μιλούμε μοναχά για τα πρότυπα στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται τα εργαστήρια αυτά και για τη διαπίστευσή τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοιόδης συγητές, συναντηθήκαμε χτες, ευχαριστώ αυτούς που ήρθαν. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση, δεν θα μπω στις πολλές λεπτομέρειες, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέματα, σε δύο ιδέες που ακούστηκαν από τους κοιόδης εισηγητές και που έχουν σαν στόχο να βελτιώσουν το κείμενο. Τώρα για το χρόνο χρονοδιάγραμμα, τι να πω, δεν έχετε μπροστά σας μια έκθεση, έχετε μπροστά σας μια πρωτοβουλία απλώς και νομίζω ότι καλύτερο είναι να προχωρήσουμε με βάση την πρωτοβουλία αν θέλετε ε, γιατί μιλάμε εδώ αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν εγκληματολογικά εργαστήρια διαφορετικής ποιότητας διαφορετικής διαφορετικών ε, που λογοδοτούν σε διαφορετικά συστήματα στα διάφορα κράτη-μέλη και που τελικά αν θέλετε δίνουν και διαφορετικά αποτελέσματα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό νομίζω και βεβαίως αυτά τα αποφασίζουν ε, τα κράτη-μέλη, αυτά αποφασίζουν ποια αποδεικτικά στοιχεία είναι θεμητά στα δικαστήρια τους. Αλλά νομίζω ότι εφόσον αν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ε, αναλύσεων στα διάφορα κράτη-μέλη δεν είναι τα ίδια, μπορεί είναι ε, πραγματικά δύσκολο να εκτιμήσουμε και τον αντίκτυπο στις δίκες που γίνονται και χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα αυτά. Οπότε έχουμε αν θέλετε και στις, ε, στην απονομή δικαιοσύνη διαφορετικά standards ε, στα διάφορα κράτη-μέλη. βεβαίω να δούμε τι στάνταρτς, τι πρότυπα υπάρχουν. Υπάρχουν τα πρότυπα ISO, τα οποία εφαρμόζονται σε κάποια εργαστήρια, σε κάποιες χώρες, αλλά όχι σε όλες. Γι' αυτό η πρωτοβουλία αυτή είναι πολύ σημαντική, γιατί θα απαιτήσει από τα εργαστήρια σε όλα τα κράτη-μέλη να έχουν τα ίδια πρότυπα, να ανταποκρίνονται στα ίδια πρότυπα. Τώρα, η δικαστική αποτίμηση των αποτελεσμάτων μπορεί να παραμείνει διαφορετική στις διάφορες χώρες, αλλά τα αποτελέσματα βγαίνουν με βάση ισότιμα αν θέλετε, ισοδύναμα ε, στάνταρτ σε όλα τα κράτη-μέλη ε, η κατάσταση είναι καλύτερη. Ε, και έτσι η απονομή της δικαιοσύνης θα γίνεται με βάση πιο επακριβείς πληροφορίες. Τα τελευταία χρόνια βεβαίως έγινε πρόοδος. Όταν ήμουν υπουργό εσωτερικών στο Ηνωμένο Βασίλειο μόλις ξεκινούσαμε με τις αναλύσεις DNA. Έκτοτε τα τελευταία πέντε χρόνια συγκεκριμένα τα πράγματα εξελίχθηκαν σημαντικά σε σχέση με το DNA και σε σχέση με τα δακτυλικά αποτυπώματα. Αυτά τα εργαστήρια πραγματικά εξελίχθηκαν σημαντικά Τώρα θα αναφέρω δύο θέματα όπου μπορεί να υπάρχουν προβλήματα βέβαια. Ένα βασικό πρόβλημα είναι η χρηματοδότηση. Σε κάποιες χώρες, ιδιαίτερα στις μικρότερες χώρες της Ευρώπης, ε, είναι σημαντική η χρηματοδότηση. Άμα πρέπει να γίνει διαπίστευση των εργαστηρίων αυτών με βάση διεθνή πρότυπα και προς το συμφέρον ολόκληρης της Ευρώπης τότε η χρηματοδότηση πρέπει να είναι επαρκής Βεβαίω αυτό εξαρτάται από τα Υπουργεία Οικονομικών δεν λέω ότι πρέπει να δώσουμε ευρωπαϊκά χρήμα κονδύλια εδώ αλλά απλώς ε, λέω ότι υπάρχει ζήτημα χρηματοδότησης. Τώρα, τι είπαν οι σκιώδες συζητητές. Συζητήσαμε το ζήτημα της ανταλλαγής πληροφοριών που θα το συζητήσουμε σε άλλα θέματα της ημερησίας διάταξης. Είναι πολύ σημαντική η ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά θα πρέπει τα στοιχεία αυτά που ανταλλάσσουμε να είναι αξιόπιστα, να είναι υψηλής ποιότητας διότι η ανταλλαγή πληροφοριών που δεν είναι ε, το ίδιο καλές ε, ή δεν είναι αξιόπιστες ε, δημιουργεί πρόβλημα και θα δημιουργήσει και πρόβλημα αν θέλετε εμπιστοσύνη στις αρχές που ανταλλάσσουν τις πληροφορίες αυτές και κάτι τι άλλο <coughs> θα ήταν ευκταίο παρόλο που οι μικρές χώρες ίσως δεν, μπορούσαν, δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν. Υπάρχει μοναχά ένα διαπιστευμένο εργαστήριο ε, πάνω από ένα διαπιστευμένο εργαστήριο από, σε κάθε χώρα με ένα και μόνο εργαστήριο στην κάθε χώρα με μια μονοπολιστική κατάσταση αν θέλετε ίσως τα πράγματα δεν θα ήταν τόσο καλά αυτά τα δύο ζητήματα λοιπόν αυτές τις δύο ιδέες ανέφερες και όλοι τις και τους ευχαριστώ για τις ε, ιδέες ε, αυτές Κύριε Πρόεδρε, είμαι υπέρ τη συζήτηση του θέματος αυτού. Δεν συμφωνώ με το χρονοδιάγραμμα. Νομίζω παρόλα αυτά ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, και να υποστηρίξουμε την έκθεση. Αλλά καθιστώ σαφέ, παρόλο που δεν βλέπω να λέγει ε, να μπορώ να το βάλω αυτό στο κείμενο, θέλω να καταστήσω απολύτω σαφέ ότι αυτό θα πρέπει να είναι απλώ το πρώτο βήμα. Περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανακάμψει με καινούριε προ... προτάσεις ιδιαίτερα για το πώς άμα φτάσουμε στην επιδιωκόμενη ποιότητα θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ποια θα είναι η χρήση των αποτελεσμάτων αυτών των εργαστηριακών αναλύσεων νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό για την προστασία του πολίτη και για την προστασία των πληροφοριών που, το, και των αποτελεσμάτων που θα προέρχονται από αυτά τα εργαστήρια που θα έχουν πλέον καλή ποιότητα και εγγυημένα standards. Ευχαριστώ κύριε Χομπ. Εκ μέρους της Προεδρίας Λίζα Μπόλιγκερ. Παρακαλώ. Thank you. Thank you. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους σας. Να ξεκινήσω Καταρχάς, ε, ευχαριστώ τον κύριο Κέρκοπ, τον εισηγητή και τους ε, σκιώδες εισηγητές για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για να σημειωθεί πρόοδος υπό τις ε, παρούσες συνθήκες. Φυσικά το εκτιμά αυτό ιδιαίτερα η Προεδρία και το Συμβούλιο. Στην παρούσα φάση, στο εσωτερικό του Συμβουλίου, νομίζω ότι τα πιο πολλά τμήματα της πρότασης πλέον έχουν αναλυθεί και έχουν συζητηθεί επαρκώς. Και είναι, υπάρχουν στοιχεία τα οποία προχωράμε πάρα πολύ καλά σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη, σε ό,τι αφορά τα κτίρια ποιότητα για τα εγκληματολογικά εργαστήρια, τα οποία θα εγκριθούν μέχρι το τέλη του έτου. Τώρα, για τα σχόλια τα οποία μόλις έκανε ο κύριος Κέρκοπ. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τα στοιχεία τα οποία έθιξε, ότι όντως θα πρέπει να αποτελέσει αυτό ένα πρώτο βήμα για να εξεταστεί η ποιότητα των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Θεωρούμε ότι είναι κατεπίγουσα σημασία να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να βελτιωθεί η ποιότητα αυτή και σε άλλους τομείς, όπως αναφέρατε, για θέματα περαιτέρω αξιοποίηση τη ε, ποιότητα αυτή σε ό,τι αφορά τι δραστηριότητε ε, εφαρμογή του νόμου. Για το τελευταίο στοιχείο που αναφέρατε, ότι θα πρέπει να υπάρχει παραπάνω από ένα διαπιστευμένο εργαστήριο ανά κράτος μέλος. Αυτό το εξετάσαμε στην πρόταση αυτή σε ό,τι αφορά τους παρόχους ε, υπηρεσιών τέτοιων που θα μπορούσαν να είναι δημόσιες υπηρεσίες. Φυσικά ένα θέμα είναι πόσες τέτοιες υπηρεσίες θα υπάρχουν, αλλά κοιτώντα, ε, για παράδειγμα το, την περίπτωση της Σουηδίας, θα διαπιστεύσουμε για παράδειγμα τα αστυνομικά εργαστήρια. Υπάρχουν 20 τέτοια εργαστήρια στη Σουηδία. Να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειές σας και ανυπομονούμε να ακούσουμε και την ε, θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σίγουρα θα αποτελέσει μια χρήσιμη συμβολή για τις συζητήσεις του ιστορικού του Συμβουλίου. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Ρενέ Φαντέικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Κέρκοπ για τα σχόλια τα οποία κάνατε σε ό,τι αφορά το θέμα για... Uh, για τη χρηματοδότηση. Για την χρηματοδότηση των εθνικών και διεθνικών προγραμμάτων. Ασφαλώς και θα προσπαθήσουμε να διαθέσουμε τα σχετικά κονδύλια για το δεύτερο θέμα. Για τη διαπίστευση πλέον του ενός ε, εργαστηρίου ανακάτως μέλλον. Συμφωνούμε με όσα είπε και η Σουδική Προεδρία και σε ό,τι αφορά το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κατά πόσο χρειάζονται περαιτέρω πρωτοβουλίες μετά την εφαρμογή της παρούσας πρωτοβουλίας, θα το εξετάσουμε. Θα δούμε κατά πόσο χρειάζονται και άλλες ε, πρωτοβουλίες μετά την εφαρμογή όμως της παρούσας ε, πρωτοβουλίας. Αυτά από την Επιτροπή. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δύο βουλευτές ζητούν το λόγο. Ο κύριος Διόγκ. Α, κι άλλοι, κι άλλοι. Όχι, δεν είναι μόνο δύο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι μάλλον σύντομος, γιατί όντω ήταν πολύ ωφέλιμη η συνάντηση με τον εισηγητή χτες και είμαι πεπισμένος ότι θα προχωρήσουμε σωστά. Πολύ λίγα στοιχεία διαφωνίας έχουμε ίσονο σημασία και συμφωνώ με όσα δήλωσε ο εισηγητή. Γιατί ζήτησε το λόγο όμω. Για να πω κάτι αναφορικά με την Προεδρία και το Συμβούλιο. Κοιτάω τα θέματα εγκληματολογικής συνεργασίας. Τι διαπιστώνω. Κάτι που με απογοητεύει και κάτι που πραγματικά είναι ανησυχητικό. Βλέπουμε πολλή συνεργασία προτού έχουν συμφωνηθεί οι δικλείδες, ε, για παράδειγμα, ε, την ποιότητα των δεδομένων. Και θέλω λοιπόν να καλέσω το Συμβούλιο και την Επιτροπή και μπορούμε να συζητήσουμε και το περιεχόμενο του προγράμματος της Στοκχόλμης να καταθέσουν ένα όραμα, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά τον σεβασμό καταρχάς των δικαιωμάτων των ε, ανθρώπων και της ποιότητας των δεδομένων. Προτού ε, γρήγορα και βεβαιασμένα, αν θέλετε, ξεκινήσουμε διάφορες μορφές συνεργασίας. Άρα, στηρίζω τον εισηγητή και καλό το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν τα θέματα αυτά και να υποβάλουν, αν θέλετε, ένα πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά. Ο κύριος Άλβαρο, ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι σκιώδης για την ε, έκθεση αυτή. Ζητώ τον λόγο γιατί στην προηγούμενη θητεία ήμουν συναρμόδιος για την ε, συνθήκη της Προύν σχετικά με τα δεδομένα αυτά. Και έχετε απόλυτο δίκιο, συνάδελφοι. Ρυθμίζουμε την ανταλλαγή δεδομένων χωρίς να ξέρουμε τι ανταλλάσσουμε ουσιαστικά. Επειδή δηλαδή υπάρχει συλλογή δεδομένων σε κάποιες χώρες, δεν σημαίνει ότι είναι ίδια η ποιότητα και ότι μπορούν αυτόματα να συγκριθούν. Θα είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει και με τον ε, ε, Επιτρόπο Μπαρό το 2007 και το 2008 στο Προύν ε, συμφωνήσαμε να εξισώνουμε τα στοιχεία DNA. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι τα δεδομένα αυτά δεν συλλέγονται μόνο με διαφορετικό τρόπο στις χώρες, δηλαδή δεν έχουμε μόνο διαφορές ε, συλλογής, αλλά έχουμε και διαφορές τεχνολογίας ε, για την επεξεργασία τους. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και γιατί επηρεάζουν ε, την κατάσταση, γιατί όταν τα συλλέγουμε αυτά τα στοιχεία, τα εξισώνουμε ουσιαστικά το ένα με το άλλο. Όπως και με τα δακτυλικά αποτυπώματα. Δεν συλλέγουμε το συνολικό δακτυλικό αποτυπώμα, Δηλαδή έχουμε κάποια ε, στοιχεία, κάποια στοιχεία σύγκρισης και αυτά ε, συγκρίνουμε. Αυτό γίνεται και με το DNA. αλλά είναι διαφορετική και η εξίσωση αν θέλετε. Υπάρχουν δύο διαδικασία. Στη μία περίπτωση, για παράδειγμα, συγκρίνουμε έξι σημεία αναφοράς για την ε, εξίσωση του DNA και στην άλλη περίπτωση έχουμε εννέα στοιχεία σύγκρισης και άμα συμπίπτουν αυτά τα νέα στοιχεία, τότε θεωρείται ότι είναι ίδιο το DNA ταυτόσιμο. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν ε, ότι υπάρχουν τρία παραπάνω στοιχεία και άρα αυτό αυξάνει την πιθανότητα ε, σφάλματος. Και να φανταστείτε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα εγκληματολογικά στοιχεία. Δηλαδή στο δικαστήριο είναι αντιαφισβήτητα αυτά τα στοιχεία. Δεν ε, μπορούν να αμφισβητηθούν. Και αν υπάρχει τέτοιο περιθώριο σφάλματος, με άλλο τρόπο δηλαδή να συλλέγονται, με άλλο τρόπο να συγκρίνονται, αυτό είναι επικίνδυνο. Και αυτά όλα είναι αντιαμφισβήτητα στα δικαστήρια. Δεν πρέπει να έχουμε δηλαδή παρόμοια πρότυπα μεταξύ των κρατών μελών, πρέπει να έχουμε τα ίδια ακριβώ πρότυπα. Θα πρέπει με τον ίδιο τρόπο να συλλέγονται, να επεξεργάζονται, να τη χάνουν επεξεργασία με τον ίδιο τρόπο και να ελέγχεται με τον ίδιο τρόπο κατά πόσο είναι ταυτόσιμα. Και γι' αυτό θα πω το εξή. Ο τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται ενώπιον του δικαστηρίου θα πρέπει και αυτό να είναι ταυτόσιμο στα διάφορα προκειμένου να υπάρχει και δικαστική ασφάλεια, αλλά και να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των ε, στοιχείων αυτών και να μην προκύψουν τραγικές ε, εσφαλμένες ε, αποφάσεις δικαστηρίων. Και νομίζω λοιπόν ότι και προς τα κράτη-μέλη και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να απευθύνουμε έκκληση προκειμένου να κάτσουμε και να σκεφτούμε πρωτού ε, αρχίσει αυτή η συνεργασία να εξασφαλίσουμε τα ίδια πρότυπα. Όχι μόνο για το DNA και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Αυτό ισχύει σε όλα τα στοιχεία των ε, βάσεων δεδομένων. Δηλαδή, να περιορίσουμε το περιθώριο σφάλματος και σε ό,τι αφορά την ταχύτητα της όλης πρότασης, νομίζω ότι ως Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να δεχτούμε να μας ασκηθεί πίεση. Φυσικά θα πρέπει να ε, προχωρήσει γρήγορα το πρόγραμμα, αλλά αν κάτι μα δίδαξαν τα τελευταία χρόνια είναι ότι πρέπει να προτιμήσουμε την ποιότητα και όχι την ταχύτητα, για να μην υπάρχουν προβλήματα αργότερα. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα πρώτα θα ήθελα να υποστηρίξω αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες Τη χτεσινή συζήτηση με τον κύριο Κίρκοπ τα συζητήσαμε τα ζητήματα αυτά και όντως συμφωνήσαμε ότι αυτά που προτείνει εδώ η Κομισιόν και το Συμβούλιο είναι σωστά. Βεβαίω στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι πάντα αξιόπιστα τα στοιχεία τα οποία ανταλλάσσονται ένα θέμα αυτό δεύτερο είναι ότι Πολλέ φορές οι αρμόδιες αρχέ στα διάφορα κράτη-μέλη που θα έπρεπε να ανταλλάσσουν τα στοιχεία αυτά δεν κάνουν την ανταλλαγή αυτή. Λοιπόν, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και τα δύο αυτά πράγματα δεν θα συμβαίνουν στο μέλλον, διότι δεν είναι σωστό. Βεβαίως, αλλά οι προτάσεις του Συμβουλίου και της Κομισιόν είναι πολύ σημαντικές για την εσωτερική ασφάλεια και για την συνεργασία των αρμόδιων αρχών στα διάφορα κράτη-μέλη, αλλά, αλλά ε, θα πρέπει να φροντίσουμε να μπορούν αυτά τα στοιχεία να είναι συγκρίσιμα και αξιόπιστα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα άλλο θέμα τώρα. Ο κύριος Κίρκοπ είπε ότι λόγω του ο, χρονοδιαγράμματος δεν υπάρχει ακόμη έκθεση, δεν υπάρχει έκθεση εκ μέρους του, δεν έχει υποβληθεί έκθεση. Οπότε τροπολογίες δεν μπορούν να υπάρχουν. Μήπως λοιπόν θα μπορούσαμε να αλλάξουμε κάποιες προθεσμίες για να μπορέσουμε να έχουμε έκθεση και κατάθεση τροπολογιών. Ευχαριστώ κύριος Μπόντ. Eh, Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο γιατί δεν συμφωνώ με τη γραμμή που παρουσιάζει το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Θεωρώ ότι η διαπίστευση των εγκληματολογικών εργαστηρίων μπορεί να καταργηθεί τελείω. Και γιατί. Γιατί δεν σημαίνει τίποτα, τίποτα σας λέω, αν τα εγκληματολογικά εργαστήρια είναι διαπιστευμένα, αν ε, τηρούν κάποια πρότυπα. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα για την ποιότητα της έρευνάς μας. Θα πρέπει να ρυθμιστούν θέματα ε, όπως για παράδειγμα η ποιότητα των ερευνών ε, στο, στα, στον τόπο του εγκλήματος. Θα έλεγα λοιπόν ότι τι αναζητούμε. Θέλουμε ένα καινούργιο κώδικα για την Ευρώπη, αλλά δεν πρόκειται να συμφωνήσω ούτε εγώ ούτε το, η ομάδα μου, το κόμμα μου. Γιατί ζητώ λοιπόν να καταργηθούν αυτές οι τακτικές ε, για να μην ε, έχουμε πολλές διάσπαρτες ρυθμίσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Δρομέδα. Γρήγορα, γρήγορα κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Κύποφ όσα μας είπε στις δεν ήμουν, αλλά δεν στο ενδιαφέρον ότι θα ήθελα σαν και ο να παρακολουθήσω το θέμα. Πρώτα απ' όλα να πω για τη διαπίστωση ότι για τη μεταφορά στοιχείων ε, θα πρέπει να είναι ορμοσμένα αυτά τα στοιχεία για τη συλλογή και στην όλη διαδικασία. Και συμμερίζουμε αυτή την ανάγκη ότι πρώτα βάζουμε τα βόδια και μετά το κάρο από πίσω ακολουθεί. Έτσι το λέμε και στην Ισπανία. Αυτή είναι η στρατηγική, είναι σίγουρη και το δεύτερο, η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με την ύπαρξη παραπάνω από ενός Ινστιτούτου. Ε, όπως στην Ισπανία, αποκεντρωμένο Ινστιτούτα ανάλογα με τις αρμοδιότητες κάθε αυτόνομης κοινότητας, περιφέρειας και το ίδιο συμβαίνει σε διάφορες χώρες. Και όσον αφορά τις αρμοδιότητες για αυτή τη διανομή. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες ακριβώς, δεν ξέρω πώς έχει κατάσταση σε όλη την Ευρώπη, αλλά πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να μπορέσει κανείς να ανταποκριθεί. Εδώ λοιπόν όταν μιλάμε για διαφορά ανάμεσα στην ε, δημόσια πτυχή ή στην ιδιωτική πτυχή σχετικά με αυτά τα αισθητούτα, τι γίνεται, είναι ρυθμισμένα αυτά, τυποποιημένα και ποιε είναι οι σχετικέ προοπτικές τώρα και για το χρονοδιάγραμμα για να καταλάβω και εγώ να ξέρω τι γίνεται ακριβώ, τι ημερομηνίε υπάρχουν για την επεξεργασία τη έκθεση αυτή. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Και τώρα, εκτός αν ε, η Σουηδική Προεδρία ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουν το λόγο, να επανέλθουμε, να ξαναδώσουμε το λόγο στον κύριο Κίρκχοπ. Θέλετε το λόγο Προεδρία, Κομισιόν, όχι. Ωραία. Ο εισηγητής τότε. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ήταν σύντομη βέβαια η συζήτηση αλλά πολύ ενδιαφέρουσα θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους ομιλητές για κάποια θέματα. Για το θέμα της εθνικής κυριαρχίας υπάρχουν πάρα πολλά πρότυπα ίζο που εφαρμόζονται διεθνώς σε πάρα πολλούς τομείς και βεβαίως όλοι μας είμαστε υπέρ της εθνικής κυριαρχίας αλλά η οθέτηση προτύπων ίζω δεν είναι ξένη επέμβαση ε, και ιδιαίτερα σε θέματα σαν και αυτό που συζητούμε χρειάζεται να έχουμε διεθνή πρότυπα και ε, που δεν είναι λόγο πρόκειται για τελεοθυρία όπως φαίνεται να πιστεύουν κάποιοι Υπάρχουν κάποια πρότυπα τώρα και ακόμη και αν εφαρμόσουμε τα διεθνή πρότυπα ε, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα για την αμοιβαία αναγνώριση, για την εκτίμηση που θα κάνουν τα κράτη-μέλη, για το, τα πρότυπα αυτά καθεαυτά και για τα αποτελέσματα άλλων εργαστηρίων και των δικών τους. Ε, δεν λέω ότι θα επιληθούν όλα τα προβλήματα. Ε, και πρέπει να δούμε πώς γίνονται οι ανταλλαγές πρώτα ε, όταν θα γίνονται οι ανταλλαγές για να δούμε αν πρέπει να διορθωθούν και άλλα πράγματα αλλά κύριε Πρόεδρε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα είναι να βάλουμε κάποιες βάσεις να έχουμε κάποια βασικά πρότυπα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν βασικά πρότυπα έχουμε κάποια πάρα πολύ καλά εργαστήρια στις, ε, στα κράτη-μέλη και σε κάποιες μικρές χώρες εξαιρετικά εργαστήρια και σε πιο μεγάλες βεβαίως αλλά πρέπει να έχουμε αυτά τα βασικά πρότυπα για να και μετά να προχωρήσουμε στο πώς θα χρησιμοποιούνται και θα ανταλλάσσονται τα στοιχεία και τα αποτελέσματα. Ο κύριος Αλβάρο έχει βεβαίως ιδιαίτερη πείρα για τα θέματα αυτά και ιδιαίτερα για τα στοιχεία DNA βεβαίω είναι περίπλοκα τα πράγματα κύριε συνάδελφε και ο, σίγουρα δεν θα είναι ε, η πλήρης λύση τα πρότυπα του Άιζο αλλά χαίρομαι για τα σχόλια που έκανε ο κύριος Σάλβαρο ιδιαίτερα επειδή είναι πεπειραμένο στο θέμα Τώρα για το χρονοδιάγραμμα πρόεδρε θα ήθελα να μου πείτε εσείς τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει. Όλοι παραπονιόμαστε για το χρονοδιάγραμμα. Ε, φαντάζομαι ότι όλοι πιστεύουμε το ίδιο ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό ήταν ε, απαράδεκτο. Ε, η έκθεση Kirkhope η οποία βρίσκεται μετέωρη αυτή τη στιγμή θα γίνει απτή γέρος σας το λέω, σας το υπόσχομαι αλλά όμως για τις τροπολογίες είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι τροπολογίες μπορούν να αναφέρονται μοναχά στην πρωτοβουλία και όχι στην έκθεση Κέρκχοπ, η οποία σας λέω ακόμη δεν υπάρχει θα ήθελα να πω ότι ελπίζω να υποβληθούν τροπολογίες να κατατεθούν οι τροπολογίε δεν ξέρω για τι ημερομηνίε πρέπει να τα αποφασίσετε εσεί κύριε Πρόεδρε παραμένω εδώ και λέω άλλο ένα μεγάλο ευχαριστώ για τι ε, ε παρεμβάσεις που έγιναν πρόεδρο. ωραία κύριε Κίρκχοπ η παρουσίαση του σχεδίου της έκθεσης είχε προγραμματιστεί για τις 4 με 5 Νοεμβρίου. Θα μπορούσε να γίνει εκεί. Στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Οπότε η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών 23 Οκτωβρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 16 Νοεμβρίου και Ολομέλεια, Ολομέλεια του Νοεμβρίου 2009. Βεβαίως ε, την ακριβή ημερομηνία δεν ξέρω. Αν συμφωνείτε με αυτό το χρονοδιάγραμμα, ευχαριστούμε. Κλείνουμε το θέμα αυτό και προχωρούμε στα θέματα 3, 4 και 5 και 6 που είναι τα θέματα που σχετίζονται με την Ευρωπόλ. Θα γίνει κοινή συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα 3, 4, 5 και 6 που σχετίζονται με την Ευρωπόλ. Η απόφαση για την Ευρωπόλ θα τεθεί σε ισχύ από 1η Πρώτου 2010 και η παλιά σύμβαση Ευρωπόλ θα είναι πλέον άκυρη. Οι προτάσεις που έχουμε στην ημερήσια διάταξη είναι ουσιαστικά συμπληρωματικά ή εφαρμοστικά μέτρα της απόφασης του Συμβουλίου ούτως ώστε η Ευρωπόλ να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά στο νέο νομικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται. Κάτι τι άλλο που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι επίκειται η θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας πράγμα που αλλάζει το νομικό πλαίσιο άρα και αυτό το νομικό πλαίσιο της Ευρωπόλου. σαν μέλη της ε, Επιτροπής ε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας και ιδιαίτερα ο το τέος της τη αυτή μέρα ότι όταν υιοθετήθηκε η απόφαση για την Ευρωπόλ ζητήσαμε αμέσως μετά τη θέση ισχύ της συνθήκης να μπορέσουν να γίνουν κάποιες αλλαγές και είπαμε ότι πρέπει να διευθετηθούν θέματα κυρίως και σε σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια και για την προστασία των δεδομένων, για τη διαφάνεια κτλ. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να ακούσουμε την Προεδρία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά τα μέλη της Επιτροπής μας για όλα αυτά τα τέσσερα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Να σας πω ότι το σημείο 3 κανόνες εφαρμογής που διέπουν τη σχέση της Ευρωπόλου με τους εταίρους συμπεριλαμβανομένης και της ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων και διαβαθμισμένων πληροφοριών για το θέμα αυτό η συγκήτρια είναι η κυρία Σοφία Ιντβέλτ για το 4 είναι και πάλι ο κύριος Κύρκοπης ηγητής για το απόρριτο για το σημείο 5 για τα αρχεία προς ανάλυση της Ευρωπόλ ο κύριος Διαυτεμέρα είναι εισηγητής και για το κατάλογο των τρίτων χωρών και οργανισμών με τους οποίους θα συνάψει συμφωνίες η Ευρωπόλ εισηγητής ήταν ο κύριος Γιάνν Φιλιπ Αλμπρέχτ α ακούσουμε όμω πρώτα τη Σουηδική Προεδρία, τον κύριο Σόρεν Κέρτεν. Έχετε το λόγο. Yes, Mrs. Ναι, κυρία Ιντφέλτ. Ναι, πριν αρχίσουμε. λέει η κυρία Σοφία Ιντβελτ, θα ήθελα να ζητήσω από το Συμβούλιο στην εισαγωγή του, του τουλάχιστον να αναφερθεί και στις προθεσμίες οι οποίες ήταν ιδιαίτερα σύντομες. Είναι σοβαρό πρόβλημα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλει να υπομειστεί τις ευθύνε του και να εργαστεί γρήγορα. Ανέκαθεν ναι, ανταποκρινόμαστε, αλλά όταν πρόκειται για τόσο σοβαρά θέματα θεωρώ απαράδεκτες τις σύντομες προθεσμίες που επιβάλλει το Συμβούλιο. Γιατί δεν μας έδωσε περισσότερο χρόνο το Συμβούλιο. Μήπως μπορεί τώρα να, μας, να κάνει κάποιες αλλαγές και να έχουμε χρόνο τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβρη. Ευχαριστώ πολύ. Η Σουηδική Προεδρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σχετικά με τις προθεσμίες αυτές που είναι τόσο κοντινές με την παρατήρηση αυτή θα ήθελα να σας πω ότι υπέβαλα το ερώτημα και νομίζω ότι έχουν ληφθεί αρκετές αποφάσεις και το Συμβούλιο να εγκρίνει και οριστικά το θέμα. Ίσως λοιπόν από πλευρά Συμβουλίου θα μπορούσαμε να βοηθηθούμε πάνω σε αυτό. Για πιο γενική άποψη από πλευρά της Σουηδικής προθεσμία, για το χρονοδιάγραμμα. Όπως το είπε και ο Πρόεδρος, αυτό θα μπει στη θέση της ε, Συμφωνίας Europol από την 1η Ιανουαρίου του 2010. Έχουμε μέχρι τώρα διάφορες προτάσεις ε, μπροστά μας ε, και είναι από τα μέτρα που κρίνονται απαραίτητα ώστε αυτές, ε, αυτή η απόφαση Συμβουλίου να συγκεκριμενοποιηθεί. Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα είδαμε ότι όταν ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας ε, για το θέμα της ε, Ευρωπόλ σημειώθηκε ένα πρόβλημα σχετικά με αυτή τη συμφωνία για τις τροπολογίες, για τις τροποποιήσεις ε, που χρειάζονται πολύ χρονικό διάστημα γιατί στη συνέχεια θα πρέπει να επικυρωθούν σε κάθε κράτος μέλος. Ισχύουν τρία πρωτόκολλα και έχει μεταβληθεί και στο παρελθόν ε, η Συμφωνία Ευρωπόλ. Αυτό ισχύει εδώ και πολλά χρόνια και τώρα περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου τα δε μελη μαζί με την Ευρωπόλ νομίζω ότι επετέλεσαν σπουδαία εργασία για να σεβαστούν τις προθεσμίες. Και πρέπει να γίνεται αυτό για να μπορέσει η Ευρωπόλ να κινηθεί, να εργαστεί σε αυτό το νέο νομικό πλαίσιο και όπως διαπιστώθηκε και μέσω της συνθήκης της Λισαβόνας θα έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό καινούριο νομικό πλαίσιο ακριβώς για την Ευρωπόλ. Χρειάζεται να δούμε τον προγραμματισμό μας και είπαμε ότι σας ε, είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα αλλά η απόφαση του Συμβουλίου για το Ευρωπόλ θα ισχύσει από την επόμενη χρονιά. Γι' αυτό ακριβώς αυτές οι μελλοντικέ μεταβολές θα επέλθουν λαμβάνοντας υπόψη τα όσοι ισχύουν στην συνθήκη της Λισαβόνα και με τη συναπόφαση εθνικών κοινοβουλίων ε, και δεν ξέρω μήπως θα πρέπει να αρκεστώ σε αυτά εισαγωγικά ή μήπως θέλετε να κάνω συγκεκριμένα σχόλια σε κάθε συγκεκριμένη πρόταση μεμονωμένα. Νομίζω ότι αρκούν αυτά εισαγωγικά. Να περάσουμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Βιτόρια τωρα στην ευρωπαικη επιτροπη η κυρια βετορια μιτσι Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, αναμένουμε να μπούμε σε μια νέα εποχή διαθεσμικής συνεργασίας, η οποία όντως θα δώσει μεγαλύτερη δημοκρατική διάσταση στις πολιτικές που είναι βασικές για την προστασία των ε, Ευρωπαίων πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανυπομονεί να ξεκινήσει η συζήτηση για τα θέματα αυτά από κοινού με το Συμβούλιο και με το Κοινοβούλιο. Εν τω μεταξύ, έχουν ε, ληφθεί σημαντικά βήματα προς τα εμπρός με την υιοθέτηση τον Απρίλιο μια απόφασης που δημιουργεί, ιδρύει την Europol. Είναι σημαντικό να θυμηθούμε ότι το νέο καθεστώς της Europol προβλέπει μία σημαντική επισκόπηση εκ μέρους του Κοινοβουλίου στις δραστηριότητες ε, τις ε, χάρη στην διαδικασία του προϋπολογισμού αναφορικά με την Europol ως ε, καινούρια υπηρεσία. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο Και τώρα, για να ελαφρώσουμε κάπως τη συζήτηση, μάλλον να διαφωτίσουμε τη συζήτηση, να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν οι μεμονωμένοι εισηγητές. Καταρχάς, για το σημείο 3, σε ό,τι αφορά δηλαδή του κανόνε εφαρμογή που διέπουν τη σχέση τη Europol με του εταίρου, η κυρία Σοφία Ιντφέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, σε ό,τι αφορά το θέμα του χρονοδιαγράμματο. Να επανέλθω στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το Συμβούλιο για τις δηλώσεις του. Από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς προσωπικά δεν αναμειχθήκατε στην όλη διαδικασία επιλογής της ημερομηνία, αλλά πρέπει να σας πω ότι αν αυτό που λέτε είναι ότι η καθυστέρηση οφείλεται στη μεκρά διαδικασία επικύρωση των κρατών μελών και αυτό προκαλεί στα τόσο στενάχρονα διαγράμματα για το Κοινοβούλιο, νομίζω ότι το Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή δεν έχει θέσει τις σωστές προτεραιότητες και νομίζω ότι τίθεται θέμα το θέμα της επικύρωσης από τα κράτη-μέλη είναι ένα γενικότερο θέμα, το οποίο θα πρέπει να το κοιτάξουμε και σε άλλο πλαίσιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόταση που έχουμε μπροστά μας, υπάρχουν αρκετά στοιχεία τα οποία μου έκαναν εντύπωση και θα ήθελα να απαντήσω, μάλλον να λάβω απάντηση από την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά στις νομικές δικλείδες ασφαλείας και στα στοιχεία ασφάλεια των δεδομένων. Μου κάνει εντύπωση, όπω και σε πολλέ άλλε προτάσεις που έχουμε συζητήσει στο Κοινοβούλιο, ότι υπάρχουν ε, πάρα πολλά κενά, πάρα πολλά κενά, πάρα πολλοί ορισμοί οι οποίοι είναι ασαφεί. δεν υπάρχει σαφή περιορισμό του σκοπού, υπερβολικά πολλέ εξαιρέσει στου ε, κανόνε, και ο όλο σκοπό τη απόφαση είναι να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό χρειαζόμαστε. Αυτό πρέπει να έχουμε και υπόψη. Γιατί όταν, μιλάει, όταν μιλάμε για ανταλλαγή πληροφοριών, πολλέ φορέ ο κόσμο θεωρεί ότι είμαστε κατά. Όχι, όχι, αντιθέτω, εμεί είμαστε υπέρ τη ανταλλαγή πληροφοριών, δεδομένων, αλλά να υπάρχουν και επαρκείς ε, κανόνες προστασίας των δεδομένων αυτών. Και θεωρώ ότι οι προτάσει δεν πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα. Παράδειγμα, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που προτείνονται για τους κανόνες, χωρίς σαφή κριτήρια όμως που θα δικαιολογούν τις εξαιρέσεις αυτές. Για παράδειγμα, θεωρώ ότι η διατύπωση if absolutely necessary, αν είναι απόλυτα απαραίτητο, if strictly necessary, δεν νομίζω ότι αυτό είναι σαφές ε, κριτήριο, σαφώς ορισμένο κριτήριο. Ορισμοί τύπου competent authorities, αρμόδιες αρχές. Ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές. Να είμαστε Ξεκάθαρη, ποιε αρχές εννοούμε. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να διευκρινιστούν πέραν αμφιβολία Και θα ήθελα να ακούσω και την άποψη του Κοινού Εποπτικού Συμβουλίου και του EDPS για τα θέματα αυτά. Πρωτού προχωρήσουμε. Επίσης, τι μου... κάτι άλλο που με εντυπωσιάζει δεν μιλάμε μόνο για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων, μιλάμε και για την προσωπικά ε, τη μεταφορά διαβαθμισμένων εγγράφων. Και μου κάνει εντύπωση διαβάζοντα το έγγραφο ότι οι κανόνε για τη μεταφορά των εγγράφων αυτών είναι πολύ πιο αυστηροί σε σχέση με τους κανόνες για τη μεταφορά και την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων. Με άλλα λόγια, δηλαδή, προστατεύουμε καλύτερα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των κυβερνήσεων από ό,τι των πολιτών. Εδώ πέρα υπάρχει κάποια ανισορροπία, θεωρώ. Και τέλος, Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο σχόλιο, το οποίο είναι λίγο εκτός θέματος, αλλά υπάρχει μία παράγραφος η οποία αναφέρει ότι οι πληροφορίες οι οποίες έχουν ληφθεί από τρίτο κράτος μέλος με παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα πρέπει να την χάνουν επεξεργασίες. Ασφαλώς και καλωσορίζουμε την αρχή αυτή, γιατί κατά το παρελθόν στην ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν ε, τήρουταν πάντα αυτή η αρχή και νομίζω ότι αναμένουμε ακόμα εξηγήσει για τις δραστηριότητες της CIA στην Ευρώπη και τις πληροφορίες που χρησιμοποίησαν οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Τέλος, νομίζω ότι χρήσιμο θα ήταν όλοι οι συγητές και για τα τέσσερα θέματα και οι σκιώδει να συναντηθούν στο Στρασβούργο και να δούμε πώς θα προχωρήσουν. Πώς θα προχωρήσουμε το πακέτο αυτό για να εργαστούμε με ταχύτητα. Αλλά και πάλι να ζητήσω από το Συμβούλιο να μας δώσει μία αναβολή μέχρι το Δεκέμβριο. Το Συμβούλιο και αυτό θα πρέπει να εργαστεί γρήγορα, αλλά και εμεί το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε προ το συμφέρον των πολιτών. σω λοιπόν και το Συμβούλιο προ το συμφέρον των πολιτών θα μπορούσε να κάνει μια προσπάθεια τέτοια. Θέμα αξιοπιστία ε, ε, το απόρριτο του πληροφόρου τη Γκρεπόλα, κύριε Κυρκόπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με όλα όσα είπε η Σοφή. Δυστυχώ δεν μπορεί να υπάρξει πρότυπο ISO σε ό,τι αφορά το απόρριτο. Υπάρχει άιζο σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες ασφαλείας. Γι' αυτό η τελευταία συζήτηση που έγινε για τα εργαστήρια ήταν πολύ καλή και πολύ αντικειμενική. Εδώ όμως υπάρχει υποκειμενικότητα η οποία επισέρχεται. Να πω λοιπόν ότι γενικά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ε, κανόνες για τα πόρτα των πληροφοριών, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά κάποιες από τις διατυπώσεις, όπως είπε η Σοφή, είναι πολύ ασαφείς. Το άρθρο 4, για παράδειγμα, για την δημιουργία μιας νέας επιτροπής ασφαλείας και σε ποιον θα είναι υπόλογη αυτή η επιτροπή. Θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια και το προσωπικό ασφαλείας εντός της Europol. Αναφέρεται στο άρθρο 10, η επεξεργασία των πληροφοριών θα υπόκειται σε ένα βασικό επίπεδο ασφαλείας. Ωραία. Υπάρχει το βασικό επίπεδο ασφαλείας και το βελτιωμένο. Εγώ προτιμώ το βελτιωμένο προσωπικά. Και ύστερα υπάρχει το θέμα της διαβάσμησης των ε, πληροφοριών. Τα κράτη-μέλη που προμηθεύουν τις πληροφορίες θα πρέπει να είναι υπεύθυνα για τη διαβάθμιση. Ωραία, αλλά θα υπάρχει κάτι άλλο σχετικό. Περιορίζουμε τα προσωπικά δεδομένα για τα άτομα εντός ε, της Europol. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά όλα τα κράτη θα είναι σίγουρα για τις δικλείδες ασφαλείας και θα χαρούν με τις δικλείδες ασφαλείας αυτές. Και επίσης να θυμάστε ότι η Europol έχει στρατηγικούς εταίρους σε ποιο βαθμό η στρατηγική αυτή η εταίρη, δηλαδή χώρες όπως η Κολομβία, η Ρωσία, η Τουρκία και έχουμε και διαπραγματεύσεις με την Αλβανία, την Βοσνία, την την Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, την Ουκρανία και άλλες χώρες. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι στρατηγικοί εταίροι. Θα συμμετάσχουν όλοι αυτοί στη διαδικασία αυτή. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό θα είναι ασφαλές στην παρούσα φάση. Προσπαθώ, Πρόεδρε, να βοηθήσω και χαίρομαι που προχωρούμε σε θέματα απόρριτου. Αλλά θα πρέπει να σας πω ότι επί του παρόντος θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ασαφής αυτή η διαδικασία. Θα προτιμούσα να υπάρχει μεγαλύτερη βεβαιότητα και θα ήθελα, ασφαλώς και θα ήθελα να συναντηθώ και με τη Σόφη και με τους υπόλοιπους στο Στρασβούργο να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Πάμε στο επόμενο θέμα για τους κανόνες εφαρμογής για τα αρχεία δεδομένου εργασία προ ανάλυση τη Ευρωπόλ, ο κύριο Δία Τεμέρα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να κάνω ορισμένε σκέψει γενικού χαρακτήρα ξεκινώντα, Θα το γνωρίζετε όσοι ήταν εδώ παρόντε και στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Ήμουν εισηγητή ε, για το αυτό που λήφθηκε σαν απόφαση και θα εφαρμοστεί, θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου και δεν είμαι καθόλου μα καθόλου ικανοποιημένος με την απάντηση του Συμβουλίου στην πρόταση που υπευλήθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλαμε περισσότερο κοινοβούλιο, περισσότερο έλεγχο κοινοβουλευτικό και αυτό που πετύχαμε τελικά ήταν λιγότερο κοινοβούλιο, λιγότερος κοινοβουλευτικός έλεγχος. Εδώ η Επιτροπή τι λέει, ότι έχουμε τον ε, κοινοβουλευτικό έλεγχο σύμφωνα με τον προϋπολογισμό. Όχι, να σας πω ότι βέβαια έχουμε δυνατότητα συναπόφασης ε, αλλά αυτό που θέλαμε, θυμηθείτε το, είναι μαζί ας πούμε με το Κοινοβούλιο να αποφασίζεται για το διορισμό του Διευθυντού και περισσότερο πρωταγωνιστικό ρόλο του Κοινοβουλίου αλλά μας έβγαλε από τη μέση με το άρθρο 48 της απόφασης που λέει ακριβώς το εξής. Λοιπόν, τι λέει η Προεδρία του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθυντής θα εμφανιστούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφού το ζητήσει το Κοινοβούλιο για τη συζήτηση σχετικά με θέματα της Ευρωπόλ και σύμφωνα και με τους ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με την εμπιστευτικότητα το απόρριτο. Έτσι, ουσιαστικά δηλαδή μηδέν γενικά πράγματα. Πολύ λιγότερα από ό,τι συμβαίνουν στα εθνικά κοινοβούλια. Εδώ οι υπηρεσίε ασφαλεία εμφανίζονται και εμφανίζονται ελεύθερα έτσι και εδώ δεν γίνεται αυτό. Ε, συμφωνώ με τον Τίμωθη και τη Σοφία που λένε ότι εδώ έχουμε αυτά τα όρια, αυτές τις ημερομηνίε. Τι γίνεται. Αυτό το τη δέσμη Ευρωπόλ, γιατί να μην το όπως πρέπει σε μια τόσο σημαντική περίπτωση. Εδώ ε, πρόκειται για κάτι παραπάνω. Υιοθετούμε τώρα αποφάσεις για να μην υιοθετούμε αποφάσεις όταν θα υιοθετηθεί, θα εφαρμοστεί η συνθήκη της Λισαβόνας. Εγώ είμαι υπέρ της συνάντησης αυτή που προτείνει η Σοφία, ώστε μαζί όλοι όσοι ενδιαφέρονται οι συγητές, οι να μπορέσουμε να θετήσουμε μια απόφαση με συνένεση από την Επιτροπή μας και συνέχεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να τα εξετάσουμε αυτά τα θέματα δε όντως και με ηρεμία. Δεν μας ικανοποιούν αυτές οι ασαφέστατες εξηγήσεις του Συμβουλίου και ακόμα λιγότερο με ικανοποιούν οι εξηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μιλάει για τη σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου στο έλεγχο μέσω του προπολογισμού και μόνο. Δεν, δεν με ικανοποιεί, επαναλαμβάνω αυτό, δεν είναι το κατάλληλο. Σχετικά τώρα με τη δικιά μου την έκθεση, Μη σας ε, κουράσω, θα πρέπει να πω πολλά. Θα χρειαστεί να μιλήσω και πολύ λοιπόν ίσως. Σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό είναι το άρθρο 14 της απόφασης να ληφθεί υπόψη που δίνει τη δυνατότητα για τη διαβούλευση αυτή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διαφορετικά σε περίπτωση συναπόφασης θα ήταν θα πρέπει να λυθεί υπόψη και το άρθρο 59.1 του Β που μιλάει πως ε, θα, τι ρυθμίσεις θα ισχύσουν για τα δελτία ανάλυσης και ακόμα κύριε Πρόεδρα σας πω ότι το περιεχόμενο της πρότασης που αναφέρεται σε γενικές αρχές για τη μεταβίβαση στοιχείων, το είδος στοιχείων, ε, προθεσμίες, συμμετοχή τρίτων, τεχνικές προδιαγραφές ακριβώς για την ταξινόμηση στοιχείων κλπ. Υπερτεχνική αυτή η πτυχή είναι, πρέπει να δούμε και την διάσταση, την πολιτική που έχει να κάνει με αυτήν την ε, μεταβίβαση, αποθήκευση χρησιμοποίηση αυτών των στοιχείων και για αυτά τα δελτία ανάλυσης και με ένα αρχείο ακριβώς ε, τη διαβούλευση, την, ε, πώς θα προσφέρει σε αυτά τα στοιχεία, τις ρυθμίσεις για τη χρησιμοποίηση και διατήρηση και διαφορετική, κατά διαφορετική αρχεία τι θα γίνει και πώς θα έχω τεχνικά μέσα για την επεξεργασία όλων αυτών. Εδώ μας έχει κόψει τα πάντα και είναι και βιαστικά σε αυτή την πρόταση για αυτή το Ευρωπόλ και που προβλέπεται ότι το Ινστιτούτο θα εργαζεται με προσωπικά στοιχεία με μόνο στόχο να ερευνά για εγκλήματα τα οποία υποπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τέλος τώρα πάμε στο τελικό, στο άλλο θέμα των τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους θα συνάψει συμφωνίες η Ευρωπόλ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, όπως είπαν και οι άλλοι συγητές, πραγματικά βλέπω και εγώ ένα πρόβλημα χρονοδιαγράμματος δεν βλέπω γιατί επήγουν όλα αυτά τα πράγματα που σχετίζονται με την Ευρωπόλ πριν τεθεί σε ισχύ που πρόκειται να τεθεί η συνθήκη της Λισαβόνας ποιος ε, γιατί βιαζόμαστε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις εδώ για την Ευρωπόλ νομίζω ότι είναι πρόωρο αν θέλετε να πάρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τέτοιες αποφάσεις διότι μετά την συνθήκη της Λισαβόνας θα υπάρχει συναπόφαση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι λοιπόν απαραίτητο να πάρθουν επιγόντως οι αποφάσεις αυτές και αυτό είναι κακό το χρονοδιάγραμμα και ρωτώ τώρα στο θέμα μάλλον το δικό μου για τα τρίτα κράτη και τους οργανισμούς με τους οποίους θα συνάψει συμφωνίες η Ευρωπόλ εδώ υπάρχουν τεράστια θέματα για συζήτηση ε, διότι πρόκειται για ανταλλαγή πληροφοριών σε ποια σε ποιε τρίτε χώρε θα δοθούν στοιχεία από τα κράτη-μέλη. Δίνω το παράδειγμα του SWIFT δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω. Ε, είναι σοβαρά τα θέματα, ευαίσθητα, λεπτά. Ε, χρόνος συζήτησης δεν υπάρχει, οπότε εμείς σαν εισηγητές και οι εισηγητές θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προθεσμίες αυτές ή αν θέλουμε αναβολή για αργότερα ή αν περιμένουμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα μετά το Δεκέμβριο ή μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πρόεδρος Βεβαίως βλέπουμε ότι όλοι οι συγητές ήταν υπερβολικά ευθύς για το θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχουν βουλευτές που θέλουν τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Yes, Mr. Arbaro, please. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. περίμενα να μου δώσετε το λόγο για να μην το πάρω μόνος μου. Άκουσα τέλος πάντων τις παρεμβάσεις των ε, εισηγητών και νομίζω ότι υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία είναι πολύ βασικά και τα οποία πρέπει να κουβεντιάσουμε. Μετά από πέντε χρόνια ως μέλος της Επιτροπής αυτής και μετά από πολλές συζητήσεις με τους συναδέλφους θεωρώ το πρόβλημα των χρονοδιαγραμμάτων ως déjà vu κάθε φορά γίνεται το ίδιο πράγμα. Αυτή τη στιγμή φταίει η συνθήκη της Λισαβόνας, άλλες φορές κάτι άλλο, αλλά πάντα πρέπει να ε, δουλεύουμε πάντα πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ήταν το δικό μου το τηλέφωνο αυτό. Λοιπόν, ε, θέλω να ρωτήσω ορισμένα πράγματα. Αυτή τη στιγμή τι, ε, τι γίνεται για την προστασία των δεδομένων τι γνώμη έχει πα, πάρει θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άρθρο 29 ε, πρέπει να το συζητήσουμε τα θέματα αυτά και να δούμε τα θέματα αυτά της Ευρωπόλ μέσα στο γενικότερο τους πλαίσιο. Πρόκειται για θεμελιώδη συζητήσεις που πρέπει να γίνουν. Τα τελευταία χρόνια πάρθηκαν κάποια μέτρα ε, ο κύριος Κοέλιο ασχολήθηκε με τα μεγάλα πληροφοριακά συστήματα και τις μεγάλες βάσεις δεδομένων. Βλέπουμε ότι θα δημιουργηθεί ένας νέος οργανισμός τώρα για το SIS2, το VIS και το Eurodac. Ένα τεράστιος οργανισμός με ε, δεδομένα. Τι θα γίνουν τα δεδομένα αυτά. Η Ευρωπόλ έχει τις δικές της βάσεις δεδομένων. Αναρωτιέμαι λοιπόν το Συμβούλιο και η Κομισιόν γιατί δεν μπορούν να μας πούν για τους διάφορους οργανισμούς που υπάρχουν ποιοι κανόνες εφαρμογής υφίστανται είναι διαφορετικοί είναι οι ίδιοι από εκεί και πέρα υπάρχει ένα θέμα εμπιστοσύνη. Δεν θέλουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, παίρνει θέσει οι οποίε να δημιουργούν προβλήματα και θυμάμαι τη συζήτηση που κάναμε για το Eurodac και για το Ευρωπολ και μας είχαν υποσχεθεί ορισμένα ε, πράγματα ότι ας πούμε τα στοιχεία του Eurodac δεν θα τα διαπραγματεύεται, δεν θα τα επεξεργάζεται η Europol. Έκτοτε αλλάζουν τα πράγματα, τροποποιούνται. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν πιο εύκολο δεζαβίου πάλι γιατί το έχουμε πει και στο παρελθόν πιο εύκολο να γίνεται μια πραγματική συζήτηση προκατακτική, μεγάλη όμως συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως είπε και η Σοφία, εμείς δεν είμαστε κατά της ανταλλαγής δεδομένων και έχουμε κάθε συνέστηση του γεγονότος ότι οι διάφορες προεδρίες του εξαμεινό προσπαθούν να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα μπορούν και η Κομισιόν πρέπει να κάνει ε, προτάσεις. Αλλά και, και εμείς δεν εξελέγημεν για να πίνουμε καφέ στι Βρυξέλλες και εμείς θα κάνουμε σωστά τη δουλειά μας ε, και προηγούμενα για, τα, για τις διαπιστεύσεις των εργαστηρίων ή ορισμένα πράγματα που ισχύουν και για το θέμα που συζητούμε τώρα θέλουμε χρόνο δεν μπορούμε μονίμως τρέχοντας ε, να προσπαθούμε να γνωμοδοτήσουμε δεν έχει νόημα δεν είναι σωστός τρόπος εργασίας αυτός και γι' αυτό και ακούσατε και τις εκκλήσεις όλων των εισηγητών που ζητούν παραπάνω χρόνο. Θέλουμε να μας δώσετε παραπάνω χρόνο. Ξέρουμε ότι για τις διαβουλεύσεις προβλέπονται μόνο τρεις μήνες κλπ. Όμως το Συμβουλίο θα έπρεπε να είναι ευέλικτο και να μπορέσει να δώσει κάποιες αναβολές. Υπάρχει το άρθρο 10, στο χρησιμοποιήσουμε λογικά. Εγώ προσωπικά έχω κουραστεί να ε, επαναλαμβάνω ότι θέλουμε να συνεργαζόμαστε αλλά η, δεν είναι μονόδρομος η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει όλοι να κάνουν τη δουλειά τους σωστά θέλουμε περισσότερο χρόνο κρίμα πρέπει να το επαναλαμβάνουμε αλλά θέλουμε αναβολή για τα θέματα αυτά Thank you, Mr. Um, Ευχαριστώ Πρόεδρε δεν ήταν εδώ οι σκιώδεις, αλλά σίγουρα θα συμμετάσχουν με τους εισηγητές. Να κάνω κάποια σχόλια εξ ονόματος της ομάδας μου. Είπατε ότι οι εισηγητές ε, είναι πολύ άμεση. Και υπάρχει λόγος. Είπε ο Αλεξάνδρ Ντεζαβού τρεις φορές. Συμφωνώ. Ο λόγος είναι ότι οι συνάδελφοι αυτοί θα πρέπει να ξέρουν ότι η ουσία της Europol είναι η τελαγή πληροφοριών. Δεν είναι μια ε, οργάνωση εφαρμογής, εκτέλεσης αν θέλετε. Το θέμα είναι να ανταλλάσσονται πληροφορίες σωστές με τους εταίρους. Όχι μόνο να διασφαλίζουμε ότι υπάρχουν απόρτες πληροφορίες, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά να διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αξιόπιστες για να καταπολεμήσουμε το έγκλημα διασυνοριακά με αποτελεσματικό τρόπο επί σειρά ετών ε, αγωνιστήκαμε προς αυτό το σκοπό και έχω ασχοληθεί με πολλά τέτοια θέματα. Η κοινοβουλευτικός λοιπόν έλεγχος είναι πάρα πολύ σημαντικός για τα θέματα αυτά και η προστασία δεδομένων είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι, είναι το α και το ω. Και αν είναι λοιπόν έτσι τα πράγματα, δεν μπορούμε να, συνε... να συνεχίσουμε με τέτοιους ορισμούς όπως αυτούς που ανέφερε η Σόφη. Απόλυτος απαραίτητο για παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς ορισμοί για το τι είναι η αρμόδια αρχή και ο κύριος Διαθεμέρα δεν ήθελε να υπησέλθει σε λεπτομέρειες, αλλά για να είμαι ειλικρινής, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες στο σημείο αυτό, γιατί μιλάμε για σημαντικές πληροφορίες για κλιματικές δραστηριότητες και όλα αυτά θα πρέπει να είναι ακριβή στοιχεία. Αυτό κάνει η Europol. Αλλά από πλευρά μα συμφωνούμε απόλυτα με τον εισηγητέ και με την απογοήτευσή του για τα θέματα αυτά και θα συμμετάσχουμε μαζί τους στην όλη διαδικασία, όπως συμμετείχαμε και στα άλλα θέματα και στις άλλες διαδικασίες για την Europol για να διασφαλίσουμε ότι η ανταλλαγή των πληροφοριών, οι καλές σχέσεις μεταξύ των εταίρων θα διασφαλιστούν. Γιατί εκεί κρύβεται η ουσία των θεμάτων αυτών. Και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει το χρόνο για να τα διασφαλίσει όλα αυτά. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, η κυρία Παδοπούλου. Δεν έχετε μικρόφωνο. The mic, please. Not working now. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα μιλήσω στο ίδιο μήκο κύματο. Θεωρώ ότι είναι πολύ εύστοχε όλε οι επισημάσει που έχουν γίνει από του προλαλήσαντε ομιλητέ και συμμερίζομαι πλήρω τι ανησυχίε για τα στενά χρονοδιαγράμματα. Τα θέματα που συζητούμε είναι νευραλγική σημασία για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Άλπρεχτ ότι δεν αντιλαμβάνομαι γιατί αυτή η βιασύνη τώρα εφόσον με την έγκριση της ηθίκης της Λισαβόνας πολλά θα αλλάξουν. Ε, επίσης συμμερίζομαι με αυτό που έχει δηλώσει ο κύριος Μωράες ότι χρειάζονται καλές σχέσεις μεταξύ των, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διαφόρων στρατηγικών εταίρων και πρέπει στον προβληματισμό που αναπτύχθηκε για τις τρίτες ε, χώρες και τη συνεργασία που πρέπει να υπάρχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση να πω και τη δική μας ανησυχία γιατί προέρχομαι από την Κύπρο και όπως πολύ καλά γνωρίζετε δεν υπάρχει αμοιβαιότητα όσον αφορά ανταλλαγή πληροφοριών σε αρκετούς τομείς στην αστυνομική παραδείγματο χάρη δικαστική συνεργασία ενώ η Interpol προσπαθεί να συνεργαστεί η Κυπριακή Αστυνομία με την Ιντερπολ, Άγκυρα, παραδείγματο χάρη, που είναι μια τρίτη χώρα η Τουρκία, δεν υπάρχει αυτή η αμοιβαιότητα. Αυτό δυσχεραίνει το έργο μα και ήθελα να θέσω ενώπιό σα ότι στον κατάλογο των τρίτων χωρών των οποίων έχω διεξέλθει, τουλάχιστον η δική μου χώρα εναντιώνεται γιατί μια από αυτές τις χώρες, η Τουρκία, και δεν εγείρω το θέμα με στόχων πολιτικών, το εγείρω απλά γιατί πρέπει να υπάρχει συνεργασία αφίδρομη. Δεν αρκεί μια χώρα μόνο να τίνει χέρι φιλίας και συνεργασίας και η άλλη να μην ανταποκρίνεται. Όταν η Ίντερπολ Λευκοσίας και η αστυνομία, η δική μα στην Κύπρο, ζητά βοήθεια από την Τουρκία, δεν υπάρχει αμοιβιότητα. Αυτό το καταγγέλλω και το έχουμε τονίσει και σε προηγούμενε ε, συναντήσεις που έχουν γίνει για το θέμα αυτό και το βάζω ενώπιό σα ζητώντας τη δική σα κατανόηση ότι η Κύπρος δεν θα πει ναι στο να συμπεριληφθεί η Τουρκία σε αυτόν τον κατάλογο των τρίτων χωρών ακριβώς γιατί δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και δεν έχει καλές σχέσεις με τις χώρες μου. Με τις άλλες τρίτες χώρες δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και εκεί οπωσδήποτε θα πρέπει η συνεργασία να αναπτυχθεί εμείς σημειώνουμε ότι η Ευρωπόλ έχει αναγνωρίσει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ανήκει στις χώρες εκείνες που ακολουθούν κατά γράμμα όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις αρχές για να ενδυναμωθεί η Ευρωπόλ, γιατί θεωρούμε ότι η ενδυνάμωσή της είναι προς το συμφέρον όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν ζητά κανείς άλλο το λόγο. Ωραία λοιπόν. Είναι σαφές ότι η όλη συζήτηση καταδεικνύει τα εξή. Καταρχάς ότι υπάρχουν έντονες αντιρρήσεις σε ό,τι αφορά την ουσία της κοινή συζήτηση ε, που λαμβάνει η χώρα, αλλά και αγανάκτηση σε ό,τι αφορά τη βιασύνη για το χρονοδιάγραμμα. Είναι λοιπόν σωστό να διοργανωθεί μια συνάντηση των σκιωδών και των εισηγητών, κατά την επόμενη Ολομέλεια στο Στρασβούργο, την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να αναδιοργανωθεί το χρονοδιάγραμμα. Γιατί το χρονοδιάγραμμα όσο έχει τώρα, να σας υπενθυμίσω ότι τι λέει παρουσίαση της, ε, παρουσία της Επιτροπής. 4 και 5 Νοεμβρίου του 2009 με προθεσμία την 6η Νοεμβρίου για τροπολογίες, 6 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, ε, ψηφοφορία στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ 16 Νοεμβρίου και ψηφοφορία στην Ολομέλεια 23 με 26 Νοεμβρίου. Αυτά προβλέπει το χρονοδιάγραμμα όσο έχει σήμερα. Αλλά θα πρέπει να αναδιοργανωθεί και υποθέτω ότι μετά από τη συνάντηση των εισηγητών και των σκιωδών θα διευκρινιστούν τα θέματα αυτά, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη ότι η απόφαση Europol θα πρέπει αναγκαστικά να τεθεί σε ισχύ από 1η Πρώτου του 2010. Άρα, για να κλείσουμε αυτή την κοινή συζήτηση, να δώσουμε και πάλι το λόγο στην Σουηδική Προεδρία και στην Ευρωπαϊκή Προεδρία. Ένα αντιδικαστικό θέμα θέλει να θέσει η κυρία Ιντσφέλτ. Ναι, προτού απαντήσει το Συμβούλιο, θα ήθελα να μας πείτε αν σκοπεύετε να διαβουλευτείτε με το κοινό συμβουλευτικό σώμα και με το EDPS. Γιατί αν σκοπεύει να πάρει τέτοιο σημαντική απόφαση το Συμβούλιο με την εμπειρογνωμοσύνη των αρμοδιοτήτων ε, προστασίας δεδομένων και επίσης να να καταλαβαίνει το Συμβούλιο ότι αυτή η διαδικασία ελέγχου δεν αποτελεί ε, ούτε μια τυπική διαδικασία ούτε μια ενόχληση. Θα πρέπει με το πνεύμα αυτό να εξετάζουμε και να θεωρούμε την διαδικασία αυτή. Να ακούσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει το Συμβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές και τους βουλευτές που παρενέβησαν και έθιξαν πολλά πολύ σημαντικά σημεία. Βέβαια, ε, πολύ γρήγορα θα έχουμε αυτές τις προθεσμίες και δυσκολεύεται το Κοινοβούλιο. Πιστεύουμε όμως ε, ότι είναι πραγματικά σημαντικό αυτό που λέει, που φρονεί το Κοινοβούλιο σχετικά. Και μπορώ να σας ε, διαβεβαιώσω ότι το Συμβούλιο θα λάβει υπόψη του τα όσα λέει το Κοινοβούλιο και προσπαθούμε να πετύχουμε μία ισορροπία γιατί όπως είπαν ορισμένοι εδώ ο στόχος των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και θα πρέπει αυτό να ρυθμιστεί και μάλιστα με σίγουρο τρόπο και με έναν δημοκρατικό έλεγχο. Όπως σας το είπα, εγώ σημειώνω προσεκτικά τις παρατηρήσεις σας, αλλά σήμερα απλά και μόνο μπορώ να πω ότι ισχύει η ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου του 2010 για την απόφαση αυτή που θα πρέπει να ισχύσει αλλά με ιδιαίτερη σοβαρότητα καταγράψαμε τις παρατηρήσεις σας και κατανοούμε και τις γενικές σας ανησυχίες σχετικά με αυτό το διαδίκτυο χρονοδιάγραμμα και αυτές τις τόσο σύντομες προθεσμίες. Λυπάμαι, αλλά... Thank you. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Μίτση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακούσαμε μεγάλη προσοχή τα σχόλια των βουλευτών τα οποία και θα μεταφέρουμε στην υπηρεσία μας. Και πάλι θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλει να υπάρξει βελτιωμένη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ίσως να μην είμαι αρκετά σαφής και λυπάμαι. Μίλησα για την εποπτεία του Κοινοβουλίου επί του προϋπολογισμού της Europol συγκεκριμένα και αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι αποτελεί το τέλος, αν θέλετε, των αρμοδιοτήτων. Απλά αποτελεί μία πτυχή που καταδεικνύει ότι έχει γίνει μία πρόοδος σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Εντφέλτ. Ναι, λυπάμαι που επανέρχομαι, αλλά δεν μου απαντήσατε, δεν μου απάντησε το Συμβούλιο μάλλον στην απάντηση μου, στην ερώτησή μου. Θα διαβουλευτείτε με το EDPS και με την Κοινή Εποπτική Αρχή. Χαίρομαι με τις γενικές σας παρατηρήσεις που είναι πάρα πολύ θερμές, αλλά πολύ λυπάμαι, δεν μου αρκούν αυτά που λέτε. Ο πρόεδρος είπε προηγουμένως ότι ήμασταν πάρα πολύ ε, ντόμπροι και πάρα πολύ ευθύς και πάρα πολύ άμεση. Και ναι, όντω, θα πρέπει κανεί να είναι μαζοχιστή για να έρχεται εδώ πέρα στην επιτροπή μα. Αλλά όπω και ο κύριο Άλβαρο, είπε και ο κύριο Άλβαρο, πάντα δεν λαμβάνουμε επαρκεί απαντήσει. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχε έρθει το Συμβούλιο και μα είπε ότι θα καθυστερήσουμε τις εργασίες μας για το EUP γιατί είναι χρήσιμη συμβολή του Κοινοβουλίου και θα περιμένουμε την εφαρμογή του, της συνθήκης της Λισαβόνες. Μπορείτε να μου πείτε γιατί το Συμβούλιο θεωρεί ότι για αυτά τα θέματα είναι σημαντική η συμβολή του Κοινοβουλίου, αλλά δεν είναι σημαντική η συμβολή του Κοινοβουλίου για τα θέματα της Γυροπόλ. Και θέλω λοιπόν να μας πείτε αν θα υπάρξει αναβολή και αν όχι γιατί. Ναι, λέει ο Πρόεδρος, από ό,τι βλέπετε, αυτά, αυτή είναι η κατάσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ξέρετε ότι τον τελικό λόγο τον έχει το Κοινοβούλιο και οι βουλευτές. Ως εκ τούτου να δώσουμε το λόγο και πάλι στους συζητητές. Ο κύριος Διαδημέρα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Προ στιγμή η τελευταία μου λέξη να μην είμαι επιθετικός ούτε απέναντι στο Συμβούλιο ούτε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να είμαι όμως περιγραφικός. Το ότι δεν μπορεί να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα το Συμβούλιο δεν το συμμερίζομαι. Μπορεί να το κάνει, μπορεί να κάνει το ίδιο και με τις μεθόδους. Για το χρονοδιάγραμμα και την αλλαγή Εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο ενός μικρού κοινοβουλίου που διαβουλεύεται απλά και μόνο είναι εντάξει το Δεκέμβριο αλλά εάν είναι ένα κοινοβούλιο με δυνατότητα συναπόφασης όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα κάνουμε τη στιγμή ακριβώς που ισχύει η συνθήκη, θα ισχύσει η συνθήκη της Λισαβόνας. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε όλα αυτά πώς θα μπορούσαμε να τα κάνουμε μαζί. Εξίσουμε το Συμβούλιο. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι λογικό, γιατί τώρα εάν επιμείνουμε και πάλι και να επιμείνουμε και πάλι για αυτή τη συναπόφαση, γιατί η Ευρωπόλη είναι ένα σημαντικό θέμα και όχι μικρή σημασίας και για τις μεθόδους ίσως μία κρόαση να οργανώσουμε και να είναι και ο κύριος υπεύθυνο για τα στοιχεία αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνομιλήσουμε και να είναι και ο διευθυντής της Ευρωπόλ και του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος παρόντες. Αυτό θέλω να πω για το χρονοδιάγραμμα όπως επίσης και για τις ακολουθητές μεθόδους. Ευχαριστώ και ο πρόεδρος. Ο κύριος Άλμπρεχτ θα ήθελα να συμφωνήσω και να κάνω μια ε, ε, ε συμπλήρωση αν θέλετε διότι εδώ δημιουργεί εντύπωση ότι πρέπει μέχρι την 1η Πρώτη του 2010 να έχουν πάρθει οι αποφάσεις αυτές διότι αλλιώς δεν θα μπορεί να λειτουργήσει η Ευρωπόλ. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Ο κατάλογος των τρίτων χωρών και το πώς με τους οποίους θα συνάψει συμφωνίες η Ευρωπόλ και ε, ο τρόπος με τον οποίο θα ανταλλαγούν οι πληροφορίες δεν είναι απαραίτητο να έχουν αποφασιστεί μέχρι την 1η Πρώτη του 2010 συνεχίζω να μην <clears throat> κατανοώ γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει να λάβει υπόψη το επιτέλους το Συμβούλιο ότι υπάρχει πρόβλημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις προθεσμίες και να αρχίσουμε και δεν έχουν όλα αυτά σχέση με την 1η Πρώτου 2010. Ο κύριος Κέρκ ναι, ακούσαμε πρόεδρε από όλους και νομίζω ότι και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κατάλαβαν ότι υπάρχουν ε, προβλήματα χρονικά τουλάχιστον βεβαίως οι εκπρόσωποι τους εδώ δεν ε, μπορούν προσωπικά να πάρουν κάποια απόφαση και να μας δώσουν απάντηση Thank you. Ευχαριστώ. Ακούσαμε την άποψη των εισηγητών. Δεν θέλω να ξανανοίξει η συζήτηση, αλλά βλέπω ότι ο κ. Μωράκης θα θέλει να κάνει μια προσθήκη. Ναι, πρόεδρε, δεν θέλω να μακρηγορήσω, απλά να μην χάσουμε αυτά που είπε ο κύριος Δίας Δεμέρα για την Σακροάση. Πρότεινε μια στρατηγική. Αυτό είναι σημαντικό για τους βουλευτές που δεν έχουν ε, ζήσει, αν θέλετε, αυτή την επίπονη εργασία για την Europol ότι ένας τρόπος για να καθιερωθεί η, α, το να, να είναι υπόλογη γύρω από είναι αυτές οι ακροάσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να το συνειδητοποιεί ο κόσμος. Και κατά δεύτερον θα ήθελα να καλέσω την ε, Σόφη να συνεχίζει την ε, εκστρατεία που έχει ξεκινήσει για να εγκαθιδρύσει σωστά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρο για να ολοκληρώσουμε λοιπόν το σημείο αυτό, να προτείνω το εξή. Το Κοινοβούλιο, όπω είπα, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να παραμείνει Κοινοβούλιο, δηλαδή να είναι αυτό υπεύθυνο και τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμά του. Δεν είναι παράλογο νομίζω βάσει της προτινόμενης στρατηγικής, καταρχάς την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο, οι και οι να θέσουν ένα νέο χρονοδιάγραμμα, κάποιες από τις προτάσεις που έγιναν από τον κύριο Ντίας και από τους άλλους να ληφθούν υπόψη, γιατί νομίζω ότι οι ενστάσεις οι οποίες ε, γέρθηκαν κάτι πρέπει να σημαίνουν και για το Συμβούλιο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσετε. Αυτά λοιπόν επί του παρόντος. Αλλά θα ενημερώσουμε και όλα τα μέλη της Επιτροπής για το χρονοδιάγραμμα, το οποίο ασφαλώς και θα αλλάξει. Περνάμε τώρα στο εξή ε, στοιχείο, στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Η κυρία Μόνικα Μπενόβα έχει καταστάσει πλέον. Άρα, να συζητήσουμε πλέον το 7, μεταφορά των διαδικασιών σε ποινικέ υποθέσεις. Ξέρετε ότι η πρωτοβουλία αυτή υποβλήθηκε από την Ισπανία και τη Σουηδία για να δημιουργηθούν κοινοί κανόνες για να διευκολυνθεί η μεταφορά διαδικασιών σε ποινικέ υποθέσεις μεταξύ αρμοδίων αρχών και κρατών μελών. Το βασικό στοιχείο είναι να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες προσαγωγής ε, και δίωξης από το ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο κράτος μέλος. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο καλούνται να γνωμοδοτήσουν μέχρι 17 Σεπτεμβρίου του 2009, Δεκεμβρίου, συγγνώμη, 17 Δεκεμβρίου του 2009. Και πάλι μας υπενθυμίζεται η σημασία της εφαρμογής της συνθήκης της Λισαβόνας και του αντίκτυπου που θα έχει στην μετέπειτα διαδικασίες. Και τώρα να μας ε, μιλήσει η συγκήτρια, η κυρία Μόνικα Μπενόβα. Και μετά να ακούσουμε και το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Άρχεται η συζήτηση. Ευχαριστώ. Το ανώτατο σκοπό ε, είναι να δημιουργηθεί ένα κοινό νομικό πλαίσιο για τη μεταφορά των διαδικασιών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός και προκειμένου να ε, αυξηθεί η αποτελεσματικότητα. Η μεταφορά τώρα διαδικασιών σε ποινικέ υποθέσεις καλύπτεται από διάφορα νομικά μέσα. Το πιο σημαντικό εκ των οποίων είναι η συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την μεταφορά διαδικασιών σε ποινικέ υποθέσεις. Ωστόσο, η συνθήκη αυτή δεν έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη και αυτό οδηγεί σε προβλήματα στις μεταξύ τους σχέσεις στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν οι διαδικασίες σε ποινικέ υποθέσεις ε, σε κανένα βαθμό σε καποια κρατημέλη και το νέο νομικό μέσο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πλήρες ε, μέσο για όλα τα κράτη-μέλη όταν θα έχει αναθεωρηθεί μετά από τις τρέχουσες συζητήσεις στην ομάδα εργασίας. την, ε, με την απόφαση που προτείνεται. Υπάρχει λοιπόν η απόφαση για την, που προτείνει τη μεταφορά βάσει ενός εντύπου αίτησης μεταφοράς το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια και για μια προκαταρτική διαβούλευση. Υπάρχει το δικαίωμα των ε, συμμετεχόντων, των θυμάτων, των θητών να ενημερώνονται για την πρόθεση μεταφοράς των διαδικασιών αυτών σε ένα άλλο κράτος μέλος. Και η άμεση επαφή μεταξύ των δικαστικών αρχών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της συνεργασίας αυτής και βάσει της πρότασης το καταγγέλων κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από ένα άλλο κράτος μέλος να ξεκινήσει τη δίωξη ενός υπόπτου σε μια ποινική υπόθεση. Το κατά πόσο το άλλο κράτος μέλος έχει τέτοια αρμοδιότητα βάσει του εγχώριου δικαίου του, όμως του δικαίου του ή βάσει του άρθρου 5 της απόφασης. Το άρθρο 5 τι λέει. Λέει ότι η αρχή παραλαβής θα αποφασίσει κατά πόσο θα αποδεχθεί ή όχι το αίτημα και κατά συνέχεια, στη συνέχεια ε, θα ισχύουν κατά την εκδίκαση οι κανόνες του κράτους μέλους παραλαβής θα πρέπει να τηρούνται οι στόχοι των ποινικών υποθέσεων και έτσι τίθεται ένα κοινό νομικό πλαίσιο για τη μεταφορά των διαδικασιών σε ποινικέ υποθέσεις μεταξύ κρατών μελών και αυτό θα καταστήσει πιο αποτελεσματική και αποδοτική τη μεταφορά αυτή για να βελτιωθεί η απόδοση δικαιοσύνης για, μέσω κοινών κανόνων για το πότε και πώς η, μια δικαστική υπόθεση η οποία έχει ξεκινήσει σε ένα κράτος μέλος μπορεί να μεταφερθεί σε ένα άλλο κράτος μέλος. Οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν να επιτευχθούν από τα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Αν χρησιμοποιηθεί το μέσο αυτό που προτείνεται στην απόφαση, τα κράτη-μέλη θα, έχουν, θα διατηρήσουν τα πλήρη δικαιώματά τους. Δεν θα επεμβαίνει η Επιτροπή. Γιατί στην παρούσα φάση δεν υπάρχει μόνο μία διαδικασία για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Άρα η απόφαση θα έχει θετικό αντίκτυπο για την εφαρμογή του νόμου και για τη διεθνή δικαστική συνεργασία και σε ό,τι αφορά την προστασία και την αρρωγή προς τα θύματα εγκληματικών ενέργειών. Και είναι συμβατή η πρόταση με την αρχή της ε, επικουρικότητας επίσης είναι συμβατή με την αρχή της αναλογικότητας γιατί περιορίζεται στο ελάχιστο στο ελάχιστο απαραίτητο προκειμένου να ε, εκπληρωθούν τα πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε να πω και το εξή. Να πω δύο λόγια για το χρονοδιάγραμμα. Αρχικά, είχα ζητήσει μια αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα για την προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Θα παρουσιάσω στις 4 και 5 Νοεμβρίου την εκθεσή μου. Θα ήθελα λοιπόν η προθεσμία για την τροπολογία τροπολογιών να μεταφερθεί από τις 6 στις 13 Νοεμβρίου. Ε, οι άλλοι Βουλευτέ θα έχουν μόνο δύο μέρες μεταξύ τη παρουσίαση τη έκθεση και τη προθεσμία υποβολής τροπολογιών και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λάβει χώρα η ψηφοφορία 1η και 2 Δεκεμβρίου όπως προβλεπόταν για να γίνει δηλαδή η ψηφοφορία στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο όπως προβλεπόταν. Thank you. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Και εδώ βλέπω ότι έχουμε πρόβλημα λοιπόν με το χρονοδιάγραμμα. Ε, ο κύριος Βαλεντάν εκ μέρους της Σουηδικής Προεδρίας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Έχει περιγράψει τα πλεονεκτήματα αυτής της απόφασης ο εισηγητής. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω τίποτα περισσότερο. Όπως είπε και εισαγωγικά λοιπόν, προς στιγμή δεν υπάρχει μια κοινή ρύθμιση για παρόμοια συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Τα πράγματα είναι διαφορετικά, αν χρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία, δι, διμερείς συμφωνίες κλπ. Εδώ προσπαθούμε να έχουμε να πετύχουμε μια ρύθμιση που να εξυπηρετεί τα κράτη-μέλη. Να υπενθυμίσω ότι από το μηδέν ξεκινήσαμε με κάτι το εντελώς μα εντελώς καινούριο. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι επίσης η λέξη κλειδί σε αυτή τη συνεργασία είναι ότι μία παρόμοια μεταφορά θα πρέπει εκεί να ισχύσει μετά το πιο σωστό, ας το πούμε έτσι, δίκαιο. Εάν δύο κράτη-μέλη πούν ότι αυτή η μεταφορά αποτελεί μια βελτίωση, θα πρέπει να είναι ακριβώς το εργαλείο αυτό το κατάλληλο για να μπορέσουν να προχωρήσουν και οι δύο αρχές. Και όπως μας έχει περιγράψει ο εισηγητής, υπάρχει μια σχετική διαδικασία για όλα αυτά. Να υπενθυμίσουμε ποια είναι η αρμόδια αρχή και πώς με την Eurojust θα έρθουν σε συμφωνία αφού συζητήσουν πρώτα πώς θα έχει όλη η διαδικασία. Και το πρόβλημα είναι να ξέρουμε τι γίνεται μετά από αυτήν την μεταφορά. Και ακόμα ένα σημείο που έδειξε ο εισηγητής είναι το άρθρο 5. Ναι, πραγματικά. Μπορεί κανείς να πει ότι αυτή η μεταφορά ε, πραγματοποιείται, ίσως όμως δεν ε, διαθέτει αρμοδιότητα το ε, κράτος μέλος όπου θα γίνει η μεταφορά. Χρειάζεται λοιπόν να το εξουδετάσουμε αυτό, να το δούμε και θα πρέπει ταυτόχρονα να δούμε και τις βασικές αρχές του ποινικού δικαίου πολλών κρατών μελών. Είναι περίπλοκο το πρόβλημα και το συζητάμε ακόμα ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ελπίζει η Προεδρία να πετύχει μια λύση ανάμεσα στα κράτη-μέλη για την όλη διαχείριση αυτού του θέματος. Αλλά επαναλαμβάνουμε το πρόβλημα είναι περίπλοκο και πολλές χώρες ε, αναρωτιούνται, θέτουν ερωτηματικά γιατί είναι δύσκολα να εξακολουθώ τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει διάθεση από όλους για να πετύχουν μια κοινή λύση. Τώρα για τα υπόλοιπα σημεία. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια συμφωνία μας τα κάτι μέλη, επαναλαμβάνω. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Εύα Σταμαδιάν από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη διότι σχεδόν όλα αυτά που ήθελα να πω τα είπε η συγγήτρια. Η Κομισιόν χαιρετίζει την πρώτη παρουσίαση αυτή που έγινε από την συγγήτρια και ε, υποστηρίζουμε τον στόχο της πρότασης αυτής όπως ήδη ελέγχθη δύο φορές, όντως υπα... λείπει ένα αυτό το ο, υ... λείπει ένας κρίκος στην όλη αλυσίδα δικαστικής συνεργασίας στην Ευρώπη. Πράγματι το κομμάτι αυτό της μεταφοράς των διαδικασιών για ποινικέ υποθέσεις ε, ε, δεν διέπεται από κοινού κανόνες. Η το ULB, το Πανεπιστήμιο των Βρυξελών το 2008 ε, έκανε μια μελέτη που κατέδειξε ότι πρέπει να υπάρχει ένας κοινό μηχανισμός για τη μεταφορά αυτών των διαδικασιών ε, και βεβαίως η Κομισιόν υποστηρίζει τον ε, στόχο αυτό εάν ελπίζοντας ότι θα καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα υψηλής ποιότητας και στάνταρτ. Έχουμε μέχρι τώρα κάποιους κανόνες που ισχύουν. Ελπίζουμε να ε, επιληθεί και το ζήτημα αυτό με έναν τρόπο αποδεκτό από όλα τα κράτη-μέλη τους ώστε να γίνεται σωστή απονομή δικαιοσύνη και σωστή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών. Thank Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ανοίγει η συζήτηση για τους βουλευτές. Η κυρία Ρενάτε Βέιβερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι σκιώδης από την ομάδα Άλτε για την πρόταση αυτή. Και για να είμαι ειλικρινής, έχω την εντύπωση ότι βρίσκομαι σε μια γκρίζα ζώνη. Θυμάμαι στην περασμένη θητεία που συζητούσαμε αντίστοιχες προτάσεις οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου και της Κομισιόν ήταν ιδιαίτερα αυστηροί κρατήρι, επέμεναν για τις προτάσεις που είχαν υποβάλει, μας εξηγούσαν πράγματα, διευκρίνιζαν πράγματα. Τώρα εδώ ακούω «We need high standards». Τι θα πει αυτό, θέλω εξήγηση για το τι σημαίνει αυτό. Να ρυθμίσουμε ε, τη σχέση μεταξύ των κρατών μελών. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Θέλετε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα αγνώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ενοχλείστε από την κατάσταση που δημιουργήθηκε ζητείτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάρα πάρα πολύ σύντομα να πάρει μια θέση ενώ επίκειται η θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας ε, όπως και ο κύριος Άλβαρο έχω και εγώ το ίδιο αίσθημα déjà vu η συγκήτρια δουλεύει για να φτιάξει ένα κείμενο που σίγουρα, όχι πιθανόν, σίγουρα τη στιγμή που θα είναι έτοιμη να το υποβάλει το κείμενο αυτό οι περιστάσεις θα έχουν αλλάξει. Δεν είναι δίκαιο αυτό το κάνατε το ίδιο πράγμα και στην, ε, στο θέμα της σύγκρουσης δικαιοδοσιών ε, το κάνετε και πάλι εδώ δεν λαμβάνετε υπόψη καθόλου αυτά που έχει πει στο παρελθόν το Κοινοβούλιο όταν μιλούσαμε για τη σύγκρουση δικαιοδοσιών και για την επιλογή δικαίου εν τότε το μιλούσαμε τότε στα άρθρα 8 και 9 για τα δικαιώματα των υπόπτων, των θυμάτων, υπάρχει δυνατότητα έφεσης κλπ. Ε, αυτά τα γνωρίσατε τελείω. Λοιπόν, ρωτώ ευθέως το Συμβούλιο. Μπορεί το Συμβούλιο να μας πει ποια άρθρα εκτός του άρθρου 5 μπορούμε ακόμη να συστήσουμε ή να τροποποιήσουμε τουλάχιστον να πάρουμε μια ιδέα για το τι ε, μπορεί να γίνει και πότε τελικά μπορεί να υποβληθεί το τελικό κείμενο και πώς μπορούμε να εναρμονίσουμε όλα αυτά τα πράγματα με το χρονοπρόγραμμα του Κοινοβουλίου. Διαφορετικά συνάδελφοι, γιατί βρισκόμαστε εδώ. Πόσες φορές πρέπει να πούμε ότι για να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας πρέπει να ανασκουμποθούμε και στο τέλος ό,τι και να κάνουμε δεν παίζει ρόλο διότι το Συμβούλιο έχει τα δικά του χρονοδιαγράμματα τα οποία αγνοούν πλήρως την ύπαρξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη γνώμη του προφανώς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Eu sunt raportor uh, din partea grupului EPP pe această decizie. Uh, eu το ίδιο όπως και η κυρία Βέμπερ για το κείμενο. φαίνεται δεν είναι του κειμένου και δεν που σε είναι και η χιλιοστή φορά που γίνεται αυτό. Ο, η, η εισηγήτρια μας τα είπε αυτά λεπτομεριακά και δεν θα σας κάνω λοιπόν άλλη παρουσίαση, άλλη αναφορά σε αυτό. Απλά και μόνο θα ήθελα να μιλήσω για δύο πράγματα που κατά την άποψή μου δημιουργούν προβλήματα και ε, θα ήθελα να ακούσω και την άποψη του Συμβουλίου και της Επιτροπής αυτό. Στο άρθρο 4 λέγεται ότι είναι σημαντικό εάν τα κράτη-μέλη θέλουν να ορίσουν άλλους αρμόδιους από ότι τα δικαστήρια τότε αυτές οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν ίσες αρμοδιότητες, την ίδια δικαιοδοσία επαναλαμβάνουμε. Για την κυρία Βέμπερ, εδώ λόγω της υποχρέωσης ε, υπάρχει υποχρέωση να ενημερώνεται ο κατηγορούμενος. Γιατί εάν απαιτείται, λέγεται θα πρέπει να ενημερώνεται κατηγορούμενος. Αλλά εγώ νομίζω σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενημερώνω το κατηγορούμενος γιατί είναι μια υπόθεση που τον αφορά. Αυτό λοιπόν θα ήθελα να ακούσω και το Συμβούλιο και την Επιτροπή πάνω σε αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κουίτστρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Άκουσα την εισηγήτρια και την εκπρόσωπο της Προεδρίας να μην λέει ότι είναι ένα μέσο για μια σωστή εφαρμογή. Πάνω σε αυτό συμφωνούμε νομίζω. Είναι σημαντικό. Αλλά εδώ θα πρέπει να δούμε και τα δικαιώματα του κατηγορουμένου που διαφέρουν από τη μία χώρα στην άλλη, στα κράτη-μέλη. Χρειάζεται να υπάρξει λοιπόν ένα τουλάχιστον ελάχιστο επίπεδο αποδοχής σχετικά με τα δικαιώματα του κατηγορουμένου. Εμείς δεν είδαμε κανένα κείμενο που να αφορά αυτό. Ίσως να περιμένουμε θετικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή. Ανησυχώ όμως. Είναι σημείο πάνω στο οποίο θα ήθελα να με καθησυχάσουν να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σαφές κείμενο για τις ελάχιστες απαιτήσει, τα ελάχιστα που ισχύουν για τα δικαιώματα του κατηγορούμενου σε περίπτωση μεταφοράς και έναξη διαδικασία σε μια καινούρια χώρα. Είναι σημαντικό να γίνεται μια μεταφορά προς όλες τις χώρες με κοινά ελάχιστα που να ισχύουν σαν βάση, αλλά και εγώ είμαι νέο μέλος και όσα είπε η συνάδελφος Ρενάτε Βέμπερ είναι σημείο ακριβώς πάνω στο οποίο χρειάζεται να σκεφτούμε πολλά και διάφορα να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Χρειάζεται ένα συγκεκριμένο σαφές κείμενο και όχι μια γλώσσα γεμάτη που δημιουργεί τόσες αμφιβολίες. Θα ήθελα να τονίσω ακόμα μια φορά ότι ναι, φρονώ ότι είναι σημαντικό το σημείο θα πρέπει να μεταφέρουμε τη διαδικασία αυτή και από τη μία χώρα στην άλλη αλλά να μην ξεχνάμε ποτέ και τον κατηγορούμενο. Γι' αυτό στο μελλοντικό κείμενο θα πρέπει να υπάρχουν τα θεμελιώδη του δικαιώματα. Σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Δεν ζητάει κανείς άλλες βουλευτής το λόγο. Άρα, και ερωτήσεις αλλά και συγκεκριμένες ε, παρατηρήσεις έγιναν προς το Συμβούλιο. Άρα, να ακούσουμε το Συμβούλιο, τον κύριο Βαλεντάν για να απαντήσει στις ερωτήσεις της κυρίας Αντωνένσκου ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο μπορώ καλύτερα στις ερωτήσεις αυτές. Σίγουρα σημειώθηκαν αλλαγές, εξελίξεις από όταν το είχαμε υποβάλει αυτό το καλοκαίρι που πέρασε. Και επαναλαμβάνω σημειώθηκαν αλλαγές στο κείμενο σε σχέση με το αρχικό και τα κράτη-μέλη κατά γενικό τρόπο συμφωνούν με τις αλλαγές αυτές. Τώρα χρειάζεται να λύσουμε ένα πρόβλημα που όπως είπα και προηγμένως είναι το άρθρο 5. Ειδικότερα για τις ερωτήσεις που μου απευθύνεται για το άρθρο 4, για τις αρχές. Ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές που θα μπορούσαν να συνεργαστούν βάσει αυτού του εργαλείου. Να σας πω ότι όπως πάντα όταν μιλάει κανείς ε, για θέματα ποινικού δικαίου και συνεργασία στα κράτη-μέλη να επαναλάβω ότι είναι πολύ διαφορετικά τον από τα συστήματά μας. Σε πολλές χώρες ο αρμόδιος είναι ο εισαγγελέα, αλλού είναι η αστυνομία η αρμόδια και η αφετηρία μας ήταν ότι θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας όλα τα συστήματα των κρατών μελών, διαφορετικά δεν θα μπορούσαν ποτέ να πετύχουμε μια συμφωνία μεταξύ τους. Και συμφωνήσαμε ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μπορούσαν να ρυθμιστούν και διαφορετικά, ε, διαφορετικές αρχές με αρμοδιότητα, όπως τα δικαστήρια ή δεν ξέρω τι, κάτι άλλο. Και ακόμα για τους κατηγορούμενους και για τα θύματα. Εμείς αναγνωρίζουμε ότι το κείμενο της αρχικής πρότασης μπορεί να ειδωθεί σαν κάτι το γενικό, αλλά ενισχύθηκε όμως στη συνέχεια μετά από όσα συζητήθηκαν. Άρα λοιπόν θα υπάρχουν ε, υποχρεώσεις και δικαιώματα και είμαστε με πιο αυστηρό τρόπο για τα κράτη-μέλη να ενημερώνουν και τα θύματα και τους κατηγορούμενους και κάτι ακόμα υπάρχει ένα σημαντικότατο σημείο ότι δεν μπορεί να είναι όμως και μια απόλυτη ανάγκη, υποχρέωση, συγγνώμη, να ενημερώνονται κάποια στιγμή ίσως για την ε, όλη ασφάλεια της ε, ανάκρισης, ίσως ορισμένα πράγματα θα μπορούσαν να παραληφθούν. Λοιπόν, χρειάζεται κύριε Πρόεδρε να μπορέσουμε να πετύχουμε μια ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα και στι υποχρεώσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και ο λόγο πάλι στην κυρία Μπενόβα. Αν θα θέλετε να θυμίσετε στους βουλευτές το χρονοδιάγραμμα που προτείνετε, αν θα θέλετε να ξαναθυμίσετε το χρονοδιάγραμμα για την προθεσμία υποβολή ε, τροπολογιών και για τη ψηφοφορία εδώ και στην ε, Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και καταρχάς την κυρία Βέμπερ. για τη συνεισφορά τους. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε τι συζητάμε και πού είναι τα προβλήματα οι δυσκολίες ίσονος σημασίας μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις ε, επαφές μας με τους εκπροσώπους του Συμβουλίου. Νομίζω ότι χρειάζεται και άλλη διαβούλευση. Μία δεύτερη δυνατότητα θα ήταν να ζητηθεί πιο πολύς χρόνος για το θέμα αυτό. πολύ ευχαρίστως να συναντηθώ με τους Κιώδης, το συντομότερο δυνατόν μάλιστα, προκειμένου να ξεκινήσουμε τις εργασίες για την ενσωμάτωση και των δικών τους προτάσεων. Το Συμβούλιο αναφέρθηκε σε κάποιες χώρες και από ό,τι κατάλαβα τα βασικά προβλήματα είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Νομίζω ότι υπάρχουν λύσεις, αλλά χρειάζεται χρόνος και χρειάζεται και καλή θέληση ασφαλώς και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων. Άρα, αυτό που περιμένω από το Συμβούλιο και την Επιτροπή είναι να δείξουν μεγαλύτερη διάθεση συνεργασία και να αναλάβουν δράσει. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τα διευκρινίσαμε λοιπόν όλα αυτά για το σημείο αυτό. Να περάσουμε λοιπόν στο τελικό σημείο της, διαταξ... της διαταξής μας. Προχωρούμε στα σημεία 9 και 10 της ημερήσιας διάταξης και για τα δύο αυτά θέματα να κάνουμε κοινή συζήτηση. Ε, το πρώτο από τα δύο θέματα αναφέρεται στο σύστημα πληροφοριών του Σέγγεν και ε, στα άτομα με θεωρίες μακράς διαμονής. Το 10 αναφέρεται η κυκλοφορία των προσώπων που έχουν βίζα μακράς διαμονής. Βασιζόμαστε σε προτάσεις της Κομισιόν προφανώς. Πρόκειται για μια δέσμη προτάσεων, δύο προτάσεων μία εκ των οποίων υπόκειται στη διαδικασία συναπόφασης. Θα δώσουμε πρώτα-πρώτα λοιπόν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Σουηδικής Προεδρίας και μετά θα προχωρήσουμε τον κύριο Κοέλιο που είναι εισηγητής και για τα δύο θέματα. Ο κύριος Δεκάστερ πρώτα-πρώτα από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Euh, Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε τις δύο μας προτάσεις, θα πρέπει πρώτα απ' όλα κάτι να υπενθυμίσουμε ορισμένες βασικές αρχές που διέπουν ακριβώς τον χώρο Σέγγεν χωρίς εσωτερικά σύνορα. Για την ελευθερία αυτό το στοιχείο του χώρου Σέγγεν Όσοι προέρχονται από τρίτες χώρες που νόμιμα είναι παρόντες ε, στο έδαφος διαμένου μια χώρα έχουν το δικαίωμα να μετακινηθούν προς τις υπόλοιπες χώρες Σέγγεν από τη στιγμή που έχουν διάθεσή τους το έγγραφο που νομιμοποιεί ακριβώς την παρουσία τους ε, σε αυτό το έδαφος του πρώτου κράτου μέλους στο οποίο παραμένουν Όσοι έχουν μια βίζα Schengen που έχει εκδώσει μια χώρα από τις χώρες του Σέγγεν μπορεί να μεταβεί παντού στις υπόλοιπες χώρες Σέγγεν γιατί αναγνωρίζεται αυτή η θεώρηση αμοιβαία από όλες τις υπόλοιπες χώρες Σέγγεν. Το κεκτημένο του Σέγγεν έχει να κάνει και με την ίση αξία ανάμεσα σε μια στάδια δαιμονής και μιας θεώρησης και όποιο έχει μια άδεια διαμονής που έχει εκδώσει μια χώρα Σέγγεν με το διαβατήριό του και αυτή την άδεια διαμονή μπορεί να μετακινηθεί σε όλο το χώρο Σέγγεν για σύντομα διαστήματα παραμονή στα υπόλοιπα κράτη του χώρου Σέγγεν. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι σαφής. Δυστυχώς ε, στην καθημερινή ζωή γίναμε μάρτυρες και σημαντικών προβλημάτων γιατί αυτή η βασική αρχή δεν γίνεται πλέον σεβαστή να σε εξηγήσω με ποιο τρόπο δεν εκδίδουν στα προξενία τους ε, στο εξωτερικό άδειε διαμονής αλλά μία βίζα ε, τύπου δέλτα μακράς διαρκείας ε, και από ό,τι γίνεται συνήθως αυτή η δέλτα μακράς διαρκείας αφού πάει σε ένα στο κράτος μέλος εκεί που έχει εκδοθεί αυτή η βίζα αντικαθίσταται από μία άδεια διαμονής. Αλλά τα τελευταία αυτά χρόνια δυστυχώς όλο και περισσότερα κράτη-μέλη δεν εκδίδουν ε, λογικά σύντομα αυτή την άδεια διαμονής και ορισμένα κράτη-μέλη σε ορισμένες περιπτώσεις ε, δεν εκδίδουν πια άδειε διαμονής ε, κυρίως για, τους, ε, για όσους ε, θέλουν να παραμείνουν μέχρι και ένα χρόνο. Και αυτό τι σημαίνει τώρα. Αυτά τα άτομα που είναι πολλά, δεν είναι μερικές χιλιάδες, αλλά είναι τουλάχιστον δεκάδες χιλιάδων, αυτοί πρέπει να παραμείνουν εκεί που έχει εκδοθεί για αυτούς η Visa Delta. Δεν είναι ε, άδεια διαμονής, αλλά λοιπόν δεν είναι βίζα θεώρηση σύντομη διαρκεία και δεν του επιτρέπει να κυκλοφορήσουν αλλού, να μετακινηθούν. Άρα λοιπόν είναι άτομα άλλης εθνικότητας που είναι νόμιμα εκεί παρόντα, αλλά λόγω διοικητικών δυσκολιών δεν μπορούν να μεταβούν σε άλλες χώρες. Και ακριβώς αυτό το πρόβλημα υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, συναντάται και ακριβώς υπήρξε μια τροποποίηση στους κανόνες Σέγγεν και είχαμε τότε την δέλτα συν γάμα θεώρηση μακράς διαρκείας αλλά ταυτόχρονα και σύντομης διάρκειας άρα λοιπόν αμοιβαία αναγνώριση για την όλη κυκλοφορία και δυστυχώς αυτή η θεώρηση γάμα ίσχυε μόνο για τους τρεις πρώτους μήνες παραμονής στη χώρα αυτή και μερικές φορές από τη στιγμή που ε, σε έξι μήνες μέσα αυτή την θεώρηση ΔΕΛΤΑ από τη στιγμή που δεν μπορούσε να, την, ε, να δώσει, να εκδώσει μια ε, άδεια αυτή η ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΑΜΑ τότε έδινε τη δυνατότητα να κυκλοφορήσουν για τρεις μήνες και μετά τίποτα αδύνατον. Και γι' αυτό ακριβώ μαζί με το Κοινοβούλιο αυτή τη δέλτα συγγάμα θεώρηση ε, αυτή καταργείται από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ αυτή η σύντομη θεώρηση που υιοθετήθηκε μόλις από το Συμβούλιο και τον Απρίλιο του 2010. Οπωσδήποτε θα απαιτείται κάτι τέτοιο να το ξεπεράσουμε και να πετύχουμε μια καινούρια λύση. Να δούμε τώρα η καλύτερη λύση ποια θα ήταν τα κράτη-μέλη να πρέπει να εκδίδουν ε, μία άδεια παραμονή και η Δέλτα να γίνεται, η θεώρηση να γίνεται άδεια παραμονή, ε, τις επόμενες μόλι μόλις ε, φτάσει στο εδάφο τους ένα ε, του μάλιστα εθνικότητας. Αυτή θα ήταν και η απόλυτα καλή λύση. Δυστυχώ, όμω από ρεαλιστική πλευρά δεν είναι δυνατό κάτι τέτοιο και η πρόταση που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έκανε δε αυτό <clears throat> τον Φεβρουάριο ήταν κάτι άλλο αλλά ε, ίσως μπορέσει τελικά να λύσει το πρόβλημα πολλών ε, ξένων υπηκών που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό. Να δούμε τώρα την πονηριά σε εισαγωγικά που χρησιμοποιείται. Αυτή η δέλτα ε, οι θεωρήσεις εκδίδονται από τα κράτη μετά από ελέγχους ε, οι έλεγχοι ή οι συνήθεις που γίνονται για την έκδοση μιας άδειας ε, παραμονής με τους ελέγχους λοιπόν αυτούς και οι άλλοι μπορούν να θεωρήσουν αυτούς τους ελέγχους ότι ικανοποιούν ε, τη διάρκεια της έκδοσης μιας άδειας διαμονής που ισοδυναμεί με μια θεώρηση. Άρα λοιπόν τι γίνεται για μακράς διαρκείας θεωρήσεις να ισχύσουν τόσο ισχύουν και για τις άδειε διαμονής ε, για την ε, ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των ξανανυπικών Λοιπόν, εάν ένας ξένος υπήκος ε, με μία άδεια διαμονής μπορεί να μετακινηθεί από τη στιγμή που αυτές οι προτάσεις θα υιοθετηθούν, μπορεί να το κάνει και με μία θεώρηση μακράς διάρκειας. Ε, μέσα του κεκτημένου Σέγγεν, τα όσα απαιτούνται για τη μετακίνηση με μία άδεια διαμονής, αυτά θα ισχύσουν χωρίς ε, να μπερδευτούμε τα υπόλοιπα της θεώρησης Δέλτα. Για να δούμε τώρα με το πληροφορικό σύστημα Schengen, με τον κατάλληλο έλεγχο πριν από την έκδοση αδειδομονής, αυτός ο έλεγχος θα γίνεται και πριν από μια θεώρηση μακράς διαρκείας. Ουσιαστικά δεν είναι ότι θα ισχύσουν καινούργια ρυθμίσεις, δεν κάνουμε κάτι τέτοιο αλλά η θεώρηση δέλτα θεώρηση μακράς διάρκειας θα ισοδυναμεί με την άδεια παραμονής. Έτσι υποβάλαμε προτάσεις ε, γιατί οι νομικοί, ε, νομικές βάσεις ε, διαφέρουν. Ένα μέρος έχει να κάνει με συναπόφαση και το άλλο με την νόμιμη μετανάστευση. Το Συμβούλιο ομόφωνα θα πρέπει να αποφασίζει με πρώτερη διαβούλευση με το Κοινοβούλιο. Θα αλλάξουν όμως τα πράγματα με τη συνθήκη της Λισαβόνας έτσι κι αλλιώς σήμερα. Ισχύει η συναπόφαση για ορισμένες υποθέσεις που θα πρέπει να ρυθμιστούν. Και ακόμα κάτι τελευταίο κύριε Πρόεδρε, αυτό το κείμενο ελπίζουμε θα μπορούσε να υιοθετηθεί και μάλιστα μέχρι τον Απρίλιο του 2010. Η πρώτη λύση εδώ και μερικά χρόνια αυτή η θεώρηση ε, ΔΣ δεν θα ίσχυε πια. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Τώρα η Επιτροπή. Όχι, όχι, όχι, όχι η Σουηδική Προεδρία. Λιντμπλαντ. Κυρία Λιντμπλαντ. Yes, please, on the Swedish presidency. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τη Σουηδική Προεδρία. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό Εξετάζουμε ιδιαίτερα προσεκτικά τις δύο προτάσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία στο χώρο Σέγγεν των ατόμων τα οποία διαμένουν νόμιμα σε μια χώρα Σέγγεν. Και η πρόταση αυτή θα πρέπει να εγκριθεί για να μπορέσει να εφαρμοστεί τον επόμενο Απρίλιο του 2010 δηλαδή για να αποφύγουμε ε, δύσκολες συνθήκες ε, για όσους διαθέτουν θεώρηση μακράς διαρκείας και που μετακινούνται στο χώρο Σέγγεν. Προεδρία, εκτιμά το ότι τόσο γρήγορα αντιμετωπίστηκε το θέμα από το Κοινοβούλιο και τονίζουμε ότι έχει σημασία μια στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανάμεσα στο Συμβούλιο, επαναλαμβάνω, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό και ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο θα μπορούσε να κάνει μέχρι μέσα σε λίγους μήνες κοινά βήματα με το Κοινοβούλιο σε διάφορες ομάδες του Συμβουλίου εξετάστηκε λοιπόν το θέμα και τώρα περιμένει το Συμβούλιο την τελική θέση του Κοινοβουλίου και περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την δική σας τοποθέτηση σε αυτό το θέμα που είναι πολύ σημαντικό για μας. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστούμε και τώρα εισηγητής κύριος Κοαγιώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εδώ, σε σχέση με αυτά τα δύο σημεία, εμείς μιλάμε για μια θεώρηση μακράς διάρκειας ε, για παρασκάρι για να σπουδάσει κανείς το Πανεπιστήμιο για μία χρόνια και έχει μια θεώρηση Δέλτα και όπως είπε ο εκπρόσωπος της Επιτρόπης τελικά ζω, ζει στο Βέλγιο σαν να είναι μια φυλακή γιατί δεν μπορεί ας πούμε να πάει στην Ολλανδία να δει μια βιβλιοθήκη που υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα βιβλία για το αντικείμενο των σπουδών του ούτε και ένα Σαββατοκύριακο δεν μπορεί να πάει μέχρι τη Βαρκελόνη γιατί δεν έχει αυτή την εγγύηση για ελευθερία μετακίνησης και το κράτος μέλος ε, στο Βέλγιο αυτή τη στιγμή αυτή τη θεώρηση μακράς διαρκείας δεν την ε, ε, άλλαξε, δεν εξέδωσε ε, άδεια παραμονής. Έτσι. Λοιπόν, ορισμένα κράτη βέβαια το κάνουν και μάλιστα γρήγορα, ορισμένα αλλά όχι. Και το κοινοβούλιο δεν μπορεί να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να το κάνουν αυτό. Το ιδανικό θα ήταν αυτές οι θεωρήσεις να αντικατασταθούν από θεωρήσεις... Ε, συγγνώμη, αυτές οι θεωρήσεις να ε, αντικατασταθούν από άδειε παραμονή. Λοιπόν, είναι μια μερική λύση. Ήταν μια μερική λύση αυτές οι θεωρήσεις, η δέλτα συν γάμα και αυτό η ελεύθερη μετακίνηση τους πρώτους τρεις μήνες. Δεν λυνόταν το πρόβλημα, αλλά λυνόταν μερικός το πρόβλημα. Αυτό το γάμα σε δέλτα τώρα θα, δεν θα ισχύει πια γιατί τον Απρίλιο θα πάψει η ισχύ σε αυτόν, επαναλαμβάνω. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να μην αφήσουμε νόμιμα εγκατεστημένους στον χώρο Σέγγεν δεκάδες χιλιάδων ατόμων να τους υποχρεώσουμε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Να τους αφαιρέσουμε αυτό το δικαίωμα, το νόμιμο τους μετακίνηση. Και θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα εκδίδονται αυτές θεωρήσεις μέσω μιας πρώτερης ε, προσφυγής στα αρχεία του Σέγγεν για να δούμε ακριβώς αυτό το σύστημα και δεν είναι όμως ε, ε, άδειε για να εισέλθουν και στι υπόλοιπε χώρες εκτός Σέγγεν. Επαναλαμβάνω, κατά την άποψή μου αυτές οι προτάσεις είναι λογικέ είναι, μέλος, είναι μέρος των νέων μας αρμοδιοτήτων και νομίζουμε ότι έτσι λύνουμε προβλήματα αυτά, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και θα ήθελα να πω ότι εκτιμώ την βιασύνη της Σουηδικής Προεδρίας. Θα πρέπει να το λύσουμε τώρα, διαφορετικά από τον Απρίλιο και μετά θα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Νομίζω λοιπόν ότι καταρχάς αυτές οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί είναι έξυπνες. Δεν βλέπω κάποια άλλη πιθανή εναλλακτική λύση και μάλιστα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας με τους ε, σκιώδεις συγητές επίσης θα συναντηθούμε για μια κοινή θέση να δούμε τι θα κάνουμε με τις θεωρήσεις μακράς διαρκείας και να μην θέσουμε βέβαια σε κίνδυνο την ασφάλεια του χώρου Σέγγεν. Ταυτόχρονα όμως να μην αφαιρέσουμε αυτή την ελευθερία, να μην στερήσουμε αυτή την ελευθερία από αυτά τα άτομα, την, ελευθερία, ε, την ελεύθερη μετακίνηση. Γιατί λάβαμε πάρα πολλά παράπονα σχετικά με τον τομέα αυτό. Ευχαριστώ και τώρα από τους βουλευτές η κυρία Μπλίσκεβης Βούτε. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των σοσιαλδημοκρατών θα ήθελα να μιλήσω για την ελευθερία κυκλοφορίας. Βάσει της συντρίας που έχουμε δει, υποστηρίζουμε την πρόταση της ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα. Δεκάδες χιλιάδες άτομα τα οποία νόμιμα διαμένουν στην ε, ζώνη Σέγγεν αντιμετωπίζουν περιορισμού. Και όπως είπε και ο εισηγητή, κάποιες φορές δεν μπορούν καν να σπουδάσουν κανονικά. Δεν μπορούν να κάνουν τουρισμό εντός του χώρου Σέγγεν και υπάρχουν σοβαρά εμπόδια. Σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν καν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, γιατί σημαίνει ότι γι' αυτό θα ταξιδεύουν πολύ συχνά. Και βλέπουμε ότι αυτά τα άτομα έχουν θεωρησει μακρά διαμονής, αλλά δεν ε, τα αντικαθιστούν, δεν αντικαθιστούν με ε, άδεια διαμονής. Δεν ξέρω γιατί κάποια κρατημέλη αρνούνται να χορηγήσουν τέτοιε άδειε διαμονή. Από όσο γνωρίζω, δεν ε, θέλουν όλα τα κράτη-μέλη να εκδώσουν ε, βίζα. Τι C. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια κατάλληλη λύση. Και εγώ θα ήμουν μάλλον υπέρ μιας απόφασης προκειμένου η θεώρηση μακράς διαμονής να είναι ε, ισότιμη με την άδεια διαμονής. Αυτό θα ήταν μια λύση για τους ε, υπηκόους τρίτων χωρών. Ωστόσο, αυτό θα σημαίνει ότι θα προκύψουν πάρα πολλά θέματα και τα ανέφερε και ο συνάδελφος εισηγητής. Ενδέχεται κάποιοι από αυτούς τους ε, υπηκόους τρίτων χωρών να χρησιμοποιήσουν, να εκμεταλλευτούν αυτή τη ρύθμιση, να πάρουν τη θεώρηση μακράς διαμονής, η οποία θα είναι ισότιμη με την άδεια παραμονής, αλλά σκοπός τους να μην είναι να σπουδάσουν ή να κάνουν τουρισμό, να έχουν διαφορετικό σκοπό. Να εγκατασταθούν στην ε, ζώνη Σέγγεν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα έγγραφα που μας έχει υποβάλει λέει ότι θα ισχύουν ίδιοι όροι για τις θεωρήσεις μακάς διαμονής και για τις άδειες παραμονής. Θα πρέπει να ζητήσουμε όμως δικλείδες ασφαλείας για τη ζώνη Σέγγεν και για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Και βλέπω ότι υπάρχει κι άλλο ένα πρόβλημα το οποίο ανακύπτει. Ενδεχομένως η απόφαση αυτή να ενθαρρύνει κάποια κράτη-μέλη τα οποία αρνούνται να εκδώσουν άδειε παραμονής, να συνεχίσουν την πρακτική αυτή, να μην εκδίδουν δηλαδή άδειε παραμονής και στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να το συζητήσουμε και ίσως θα έπρεπε να υποβάλουμε μία πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συλλέξουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από όλα τα κράτη-μέλη, να τα εξετάσουμε στην Επιτροπή εδώ στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κατανοήσουμε γιατί οι θεωρήσεις, δεν εκδίδονται μάλλον θεωρήσεις ή άδειε παραμονής. Τι δικαιολογία προβάλλουν τα κράτη-μέλη. Mrs. Tack för det, Ευχαριστώ, κύριε Κοέλιο. Επε... Μας παρουσίασε τα επιχειρήματά του και συμφωνώ μαζί του, θεωρώ ότι το Συμβούλιο κατέθεσε μια αρκετά καλή πρόταση και φυσικά θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι εξασφαλίζεται στη ζώνη Σέγγεν η ελεύθερη κυκλοφορία. Είμαι μέλος ε, και της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Θα γνωμοδοτήσω, θα έχω συμβουλευτικό μάλλον ρόλο στην Επιτροπή σας. Και σημειώνω και το αίτημα της, ε, του κυρίου Κουάγη για να συνεχιστεί η συζήτηση και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κίνγκα Γκόντ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να ε, συστήσουμε τα θέματα αυτά, τα 9 και 10 της ημερησία διάταξη. Ακούσαμε από τον κύριο Κοέλιο ότι μιλούμε εδώ για φοιτητέ, σπουδαστές, που δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι αυτούς τους δεκάδες χιλιάδους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση. Αλλά δείτε Ε, δεν μέσα στο, στην, στο χώρο Σέγγεν μπορεί να βρεθεί μια λύση αρκετά σύντομη αν θέλετε ή αυτές οι σύντομες λύσεις συνιστούν και κίνδυνο ασφάλειας και πρέπει να τις προσέξουμε ακόμη πιο πολύ ε, ο κύριος ε, καταλαβαίνω κύριε πρόεδρε ποια είναι η μεγάλη σημασία των προτάσεων αυτών για την ε, κυκλοφορία, ελεύθερη κυκλοφορία των επικών τρίτων χωρών. Αλλά έχω μια απορία. Σήμερα υπάρχει διακριτική ευχαίρεια για την έκδοση άδεια παραμονής. Ε, τη διακριτική ευχαίρεια αυτή την έχουν τα κράτη-μέλη. Επίσης, αυτή τη στιγμή η θεώρηση D+C δίνει περισσότερο χρόνο στις εθνικές αρχές για να κάνουν τις έρευνές τους και ό,τι πρέπει να κάνουν για να εκδώσουν την άδεια παραμονής. Α, αλλά τους δίνει και περισσότερο χρόνο για να κάνουν και τους ελέγχους να ερευνήσουν τα πράγματα για να δουν επίσης κατά πόσον η θεώρηση μακράς διαμονής ε, έγινε σεβαστή αν θέλετε από τον υπήκο της τρίτης χώρας που την πήρε εγώ λοιπόν ρωτώ τώρα αλλάζει η κατάσταση αυτή σχετικά με τη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών να εκδώσουν την άδεια παραμονής δηλαδή δεν αποφασίζουν πια τα κράτη-μέλη για την άδεια παραμονής ευχαριστώ πολύ κυρία Κέλλερ είναι κάπως διαφορετική η προσέγγιση μας. Συμφωνούμε βεβαίως ότι οι άνθρωποι που έχουν θεωρήσει μακράς διαμονής πρέπει να μπορούν να κυκλοφορούν μέσα στο χώρο Σέγγεν. Αλλά η βλέπουμε ότι τα στοιχεία για αυτές τις θεωρίες μακράς δήμονες θα πρέπει να καταχωριστούν στο σύστημα πληροφοριών Schengen, στο ΣΥΣ. Βλέπουμε λοιπόν άλλη μια ομάδα ανθρώπων που φακελώνεται, αν μπορώ να το πω έτσι. Και όλο αυτό κάνουμε, καινούργιες ομάδες, κατηγορίες ανθρώπων συνεχώς προστίθενται που κατηγορίζονται στα συστήματα πληροφοριών και αυτό μας ενοχλεί. φοβόμαστε ότι μπορεί να υπάρχει και μη σεβασμό των αρχών προστασία δεδομένων και αυτό είναι ανησυχητικό. Ευχαριστώ πολύ. Λέει ο πρόεδρο. Α δούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριο Δεκόστερα αν έχει να πει κάτι. Ναι κύριε πρόεδρε. Υπάρχει ένα θέμα για το οποίο θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια το θέμα της διακριτικής ευχέρειας για την έκδοση αδειών παραμονής που το, την έχουν αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε εναρμονίσει το δικαίωμα εισόδου και παραμονής για κάποιες κατηγορίες φοιτητές, ε, επανένωση οικογενειών κτλ. Εκεί το δικαίωμα ε, έκδοση άδεια παραμονής το έχει το κράτος μέλος αλλά σε λογικά χρονικά διαστήματα τρεις μήνες, έξι μήνες, ένα μήνα ό,τι μπορεί να σημαίνει το εύλογο χρονικό διάστημα και υπάρχει ουσιαστικά υποχρέωση του κράτους μέλους να εκδώσει την άδεια παραμονής και οι υποχρεώσεις αυτές δεν επηρεάζονται καθόλου από την πρότασή μας. Οι υποχρεώσεις αυτές συνεχίζουν να ισχύουν για τις κατηγορίες για τις οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Όμως υπάρχουν κατηγορίες όπως οι εργαζόμενοι για τους οποίους δεν έχει γίνει ακόμη εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, και για αυτές τις κατηγορίες τα κρατη έχουν τη διακριτική ευκαιρία και παίρνουν και την απόφαση βάσει του εθνικών τους διατάξεων αν θα δώσουν την άδεια ή όχι. Ε, ενώ εμείς μιλούμε για το μέλλον και λέμε ότι αν δίνεται θεώρηση μακράς διαμονής τότε θα πρέπει να η διακριτική ευχαίρεια του κράτους να γίνει υποχρέωση έκδοση της άδεια παραμονής. Πρόεδρος, τον τελευταίο λόγο η Σουηδική Προεδρία, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Προεδρία θα ήθελε να σας ευχαριστήσει για τις παρεμβάσεις σας και τη βοήθειά σας. Μπορούμε να πούμε ότι στην εισαγωγική συζήτηση στο Συμβούλιο αρκετά κράτη-μέλη υποστήριξαν ιδιαίτερα την πρόταση της Επιτροπής. Κατανόησαν την ανάγκη που εμφανίστηκε να λυθούν παρόμοια προβλήματα και διάφορες όμως αντιπροσωπείες θέλησαν να τονίσουν και το θέμα που έχει να κάνει με την ασφάλεια τελικά και ορισμένες ε, βασίστηκαν σε αυτή την ανάγκη γιατί για να προβάλλουν ε, αντιρρήσεις γιατί από δικής τους εθνικής πλευράς ε, αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες. Το μεγαλύτερο μέρος όμως κατανόησε ότι θα πρέπει να το πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε. Κοέλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα σαφείς οι εξηγήσει της ε, και ενισχύεται έτσι η ιδέα ότι το Κοινοβούλιο το όλο θέμα για αυτές τις δύο προτάσεις το βλέπει σαν μία ενιαία δέσμη Υπάρχουν διαφορετικές αρμοδιότητες, τη μία είναι η συναπόφαση, στην άλλη στο άλλο θέμα όχι αλλά οι δύο προτάσεις αποτελούν μέλος μιας δέσμης και ακριβώς σαν ένα σύνολο θα εξεταστεί, θα αναλυθεί. Σε ό,τι αφορά το θέμα το οποίο έθεσε ο κ. Μπουζουτήλ, εν μέρει το απάντησε επαρκώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που θέλω εγώ να υπογραμμίσω είναι αυτό που έχουμε πει και στο παρελθόν είναι εν μέρη ορθό ότι η θεώρηση D C έλυσε το πρόβλημά μας, αλλά σύμφωνα με το νέο κώδικα δεντολογίας που θα εφαρμοστεί από το Απρίλιο και μετά και που εγκρίναμε στο Κοινοβούλιο, καταργείται αυτού του τύπου η θεώρηση. Δεν θα υπάρχει πλέον. Άρα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα το οποίο και θα πρέπει να επιλύσουμε με κάποια μέτρα. οι πιο πολλοί ομιλητές φαίνεται ότι συμφωνούν για τις λύσεις που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Νομίζω ότι θα πρέπει να, προστατεύσουμε το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και παράλληλα να υπογραμμίσουμε το επίπεδο της ασφάλειας. Γι' αυτό θεωρώ ότι χρειάζονται οι απαιτήσει του ΣΥΣ σε αυτές ε, της διαδικασίας τώρα είναι δυνατόν να εκδοθεί μία θεώρηση μακράς διαμονής χωρίς να ελεγχθεί στο ΣΥΣ αν το άτομο αυτό επιτρέπεται να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν αποτελεί απειλή δεν απαγορεύεται κανείς να περάσει τα σύνορά μας και ελπίζω να συνεργαστούμε σωστά με τους ε, σκιώδεις για να βρούμε καλές λύσεις. Και να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις, ε, αν είναι δυνατόν, στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν υπάρξει ομοφωνία ή συνένεση μεταξύ των σκιωδών του Συμβουλίου και της Επιτροπής, Πρόεδρε, ευχαρίστως να υπάρξει συμφωνία πρώτης ανάγνωσης για να επιταχυνθεί η διαδικασία γιατί φυσικά θα πρέπει γρήγορα να προκύψει μία απόφαση για να επιληθεί το πρόβλημα που αντιμετάζουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Γιατί θα έχουμε πρόβλημα αν το λύσουμε το θέμα μέχρι τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, κύριε Κοέλιο. Μετά από αυτά που μας είπε και ο εισηγητής, νομίζω ότι συμφωνήσαμε για το χρονοδιάγραμμα και την διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Το χρονοδιάγραμμα ε, μετά τη διαβούλευση με τους Σκιώδης και με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, ε, μάλλον θα ακολουθήσει ενημέρωση των βουλευτών της ε, Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ. Αυτά λοιπόν. Και θα ξέρετε ότι το 11, το σημείο 11 στην ημερήσια διάταξη έχει ακυρωθεί. επειδή δεν μπορούσε να έρθει ε, το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ναι, τη δικαστικό θέλετε να θέσετε, κύριε Άλβαρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ήθελα να σας διακόψω, αλλά μιας και έχει ακυρωθεί, ίσως έχουμε λίγο χρόνο και θα ήθελα να θέσω ένα θέμα για πέντε λεπτά, αν μου επιτρέπετε, αλλά δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να σας διακόψω. Το 11 στο 12, ναι, λέει ο Πρόεδρος, έχουμε τα διάφορα. Αν υπάρχουν διάφορα, ευχαρίστως. Αλλά αν υπάρχουν ε, άλλα σημεία που θέλουν να υποβάλουν οι συνάδελφοι στα διάφορα, μπορεί να μας στάσει ο χρόνος. Γιατί μπορεί να μην ολοκληρώσουμε νωρίτερα. Στα διάφορα, λοιπόν, αν θέλετε να πάρετε το λόγο, ευχαρίστω. Αλλά να είστε σύντομο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε με κάθε σεβασμό σε αυτό που είπατε να είμαι σύντομος θα προσπαθήσω να είμαι αλλά είναι ένα αρκετά σοβαρό θέμα είναι το περίφημο SWIFT και συνεχώς ακούμε πράγματα για το SWIFT υπάρχουν έγγραφα που κυκλοφορούν φαίνεται μεταξύ των κρατών μελών και που υποτίθεται ότι ενημερώνουν αλλά στην καλύτερη περίπτωση είναι χάσιμο χρόνο για να τα πω τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν ξέρω αν ξέρατε εσείς ότι τούτη τη βδομάδα ε, είχαμε πει ότι θα πρέπει να γίνει ε, η πέμπτη και τελευταία συνάντηση για το θέμα του SWIFT δεδομένων των αυτών που θα συμβούν τον Νοέμβριο.